Well, we have a long day ahead of us. So therefore we should start with the first item on the agenda, which is the vote. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο σημείο της σημερινής διάταξης, την ε, ψηφοφορία για το κοινωνικό, το καθεστώς, το κοινωνικό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διτής χρήσης. Ψηφίζουμε για την πρόταση κανονισμού και άκουσα ότι το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά χθε μεταξύ των ενδιαφερομένων και σε γενικές γραμμές υπάρχει συμφωνία για τις τροπολογίες. Οπότε θα πρέπει να ψηφίσουμε συνολικά on block για τις εξής τροπολογίες τις οποίες συμφωνήσαμε. 1, 28, 2, 3, 4, 30, με προφορική τροπολογία. 6, 7, 13, 32 με προφορική τροπολογία. 15, 16, 33, 34. Και θα σας πω στο τέλος τι απέμεινε. 17, 35, 19, 20, 36 με προφορική τροπολογία. 37, 22, 23, 38 με προφορική τροπολογία. Και την πρώτη προφορική τροπολογία. Θα ψηφίσουμε λοιπόν συνολικά on block όλες αυτές τις τροπολογίες και σε μια δεύτερη φάση θα ψηφίσουμε ξεχωριστά τις τροπολογίες 10 και 11 και έπειτα την τελική ψηφοφορία. Σωστά έχουμε πληροφορηθεί το τι συμφωνήθηκε. Could have been the same even without... Και χωρίς αυτή την ψηφοφορία το ίδιο θα είχε γίνει. Κοιτάξτε έξω. Uh, the block vote. Η ο μπλοκ ψηφοφορία λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Συμφωνήθηκε. Εγκρίθηκε. We'll check the vote against to see whether it's true or not. Θα κοιτάξουμε τις ψήφους κατά για να δούμε αν αληθεύει. Μετά, ψηφοφορία για την 10 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Συμφωνήθηκε. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ας κάνουμε έλεγχο. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Θα περιμένουμε, μην ανησυχείτε. Εψήφισαν όλοι. Προσπαθήστε να πάτε σε άλλο μηχάνημα. Everybody has voted. Εψήφισαν απαντές. Ωραία. Πέρασε. Εγκρίθηκε 18 προς 15. Τώρα ψηφοφορία για το άρθρο 11. Υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να το ελέγξουμε πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ακριβώς το αποτέλεσμα. Κύριε Πρόεδρε, έχω χάσει την κάρτα μου. Είστε υπέρ ή κατά. Υπέρ. Εντάξει λοιπόν, 19 προς 14 ψήφια. Ένας υπέρ λοιπόν και δύο επιπλέον κατά. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. να παντές. Πέρασε. Συντριπτική η έγκριση. Mm. Πρόεδρε, και πάλι υπέρ. 31 υπέρ. Ωραία λοιπόν. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο. Αφγανιστάν. Ο εισηγητής μας δεν έχει φτάσει ακόμη. Κοιτάζουμε να δούμε πού είναι.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 Because of lack of Επειδή μας λείπουν τα στρατεύματα, ο πόλεμος αναβάλλεται. Περιμένουμε τους μαχητές. Πρέπει να έρθει ο συγητής. right now. Εντάξει λοιπόν, ο ρελατόρε, ο μα μας, είναι μαζί μας. Κύριε Αρλάκη, είστε έτοιμος. Θα παρουσιάσετε την εκθεσή σας. Πρόεδρε, έτοιμος. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι η πρώτη συζήτηση Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω με συνθετικό τρόπο τη δουλειά που έκανα τον τελευταίο μήνα. Προσπαθώντας να μιλήσω για μια συνεκτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Αφγανιστάν. Το πρώτο σημείο που υπέπεσε στην προσοχή μου είναι το τεράστιο κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Αφγανιστάν μεταξύ της τρέχουσας κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης των Αφγανών αφενός και των πόρων της χώρας τα τελευταία, τα τελευταία χρόνια. Αποφάσισα λοιπόν να επισκεφθώ το Αφγανιστάν και να προσπαθήσω επιτόπου να διαπιστώσω τον αντίκτυπο της ε, διεθνούς βοήθειας στη χώρα μετά το 2001. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το βασικό πολιτικό ζήτημα, η ειρηνευτική διαδικασία στη χώρα, γιατί σχεδόν κάθε μέρα στις ειδήσει κάτι ακούμε σχετικά με το Αφγανιστάν. Άλλο ένα σημαντικό θέμα που έχει σχέση με την ειρηνευτική διαδικασία και με την ευρωπαϊκή στρατιωτική παρουσία στη χώρα είναι η κατάρτιση και εκπαίδευση της αστυνομίας στο Αφγανιστάν ώστε να υπάρξει μια πραγματική υπηρεσία ασφαλείας. Και ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα ε, όσον αφορά την Ευρώπη είναι η καλλιέργεια οπιούχων και η διακίνηση από το Αφγανιστάν προς τον ε, υπόλοιπο κόσμο. και ένας ε, συμπληρωματικός λόγος εκτός από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, ένας ε, επιπλέον λόγος ανησυχίας για το Αφγανιστάν είναι ότι η ροήνη από το Αφγανιστάν δηλητηριάζει 1,5 εκατομμύριο τοξικομανείς στην Ευρώπη. Επομένω, είναι ένα θέμα τεράστιας σημασίας για μας και θέλουμε να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα των ναρκωτικών. Για το θέμα της διεθνούς βοήθειας καταρχήν. Προσπάθησα να αξιολογήσω την κατάσταση στο Αφγανιστάν σήμερα σε σχέση με πριν από εννέα χρόνια. Ε, αλλάζει πολύ γρήγορα η κατάσταση Υπάρχει υψηλό ρυθμός ανάπτυξης για όλες ε, τις φτωχέ χώρες του κόσμου, σχεδόν όλες. Ε, από τα ταξίδια μου σε διάφορες ε, χώρες του τρίτου κόσμου, μου έχει κάνει εντύπωση το γεγονός η μεγάλη πρόοδος, κοινωνικο-οικονομική πρόοδος των λαών σε πολλά σημεία της Αφρικής και της Ασίας. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση στο Αφγανιστάν είναι ότι είδα ότι δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη ανάπτυξης. Υπάρχουν μικρές βελτιώσεις στο σύστημα εκπαίδευσης και στις υποδομές, αλλά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι οι πιο σημαντικοί δείκτες από την ε, θνησιμότητα των νεογνών μέχρι την ε, θνησιμότητα των επιτόκων γυναικών ε, μέχρι τα, τους δείκτες φτώχειας της χώρας τα τελευταία εννέα χρόνια δείχνουν ε, επιδείνωση. Όλοι αυτοί οι δείκτες. Προσδόκιμο επιβίωσης ε, μειώθηκε κατά τέσσερα χρόνια. Θνησιμότητα των ε, μητέρων στο Αφγανιστάν σκοτώνει περισσότερα άτομα από ότι ο πόλεμος. Πεθαίνουν 20.000 γυναίκες κατά τη διάρκεια του τοκετού κάθε χρόνο, λόγω έλλειψης βασικών υγειονομικών συνθήκων ενώ από τον πόλεμο σκοτώνονται 2.000 άτομα κατ' έτος. Και ο αριθμός των φτωχών στο Αφγανιστάν έχει διπλασιαστεί, αυτοί που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Η αφγανική κυβέρνηση έχει υπολογίσει ότι απαιτούνται 600 εκατομμύρια ευρώ κατέτος για την απελαγή από το πρόβλημα της φτώχειας, ώστε αυτοί που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας να φτάσουν πάνω από το όριο της φτώχειας. Η Αμερικανική κυβέρνηση δαπανά 40 εκατομμύρια ε, το χρόνο για βοήθεια στο Αφγανιστάν. Ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 ε, δισεκατομμύριο το χρόνο. Υπάρχουν και άλλοι δωρητές όπως η Ιαπωνία και άλλες χώρες. Δηλαδή υπάρχει μια ροή βοήθειας ε, που είναι περίπου 70% του ΑΕΠ του Αφγανιστάν. Πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό. Και το γεγονός ότι ο αντίκτυπος αυτή της διεθνούς βοήθειας είναι πολύ μικρός είναι η πρώτη ένδειξη που σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική πρέπει να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό το θέμα περίπου 80% της διεθνούς βοήθειας ε, που στα χαρτιά φαίνεται ότι φτάνει στο Αφγανιστάν δεν φτάνει στο, στο λαό του Αφγανιστάν και πρέπει να δούμε ποιο είναι το αίτιο γι' αυτό. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφθορά στην κυβέρνηση και στην κοινωνία του Αφγανιστάν. Και τεράστια σπατάλη στη δομή της διεθνούς ε, βοήθειας δεν ήταν τόσο σημαντικό το θέμα όταν ξεκινήσαμε την έκθεση, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες έγινε ένα καυτό ζήτημα. Το Αμερικανικό Κογκρέσο ε, την τελευταία εβδομάδα πάγωσε 5 δισεκατομμύρια βοήθειας προς το Αφγανιστάν για να μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα το πώς δαπανώνται τα χρήματα της Αμερικανικής βοήθειας ε, στο Αφγανιστάν. Και υπάρχει και μια υπηρεσία επιθεωρητών για τη βοήθεια στο Αφγανιστάν και διαπιστώνεται από τους επιθεωρητές τεράστια σπατάλη. Και η διάσκεψη του Καμπούλ, της Καμπούλ θα αντιμετωπίσει ακριβώς, ε, θα συζητήσει αυτό το θέμα και υπάρχει ε, αυτό το σημείο που πρέπει να συζητηθεί, ε, η αφγανική κυβέρνηση ζητάει να περνάει η διεθνής βοήθεια από την κυβέρνηση του Αφγανιστάν και όχι από διάφορες οργανώσεις. Έχω κάνει λοιπόν διάφορα σχόλια. Καταρχήν μας ενδιαφέρει να κατανοήσουμε την πολιτική της ευρωπαϊκής βοήθειας στο Αφγανιστάν και στην έκθεση αυτή το πιο δύσκολο ήταν να κατανοήσουμε πώς τα χρήματα τα δικά μας, τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογουμένου δαπανώνται στο Αφγανιστάν. Διότι υπάρχει μια τεράστια σύγχυση. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν κάποια συγκεντρωτική βάση δεδομένων μέσω της οποίας να μπορούν να γνωρίζουν τι δαπανούμε στη χώρα αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καλύτερα δεδομένα και τα δεδομένα αυτά ε, τα έχω στη διάθεσή μου, αλλά η γενική εικόνα είναι πολύ δύσκολο να γίνει κατανοητή. Ο αντίκτυπος ε, της ευρωπαϊκής βοήθειας προς το Αφγανιστάν ε, δεν έχει καταμετρηθεί και δεν υπάρχει τρόπος να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την παροχή βοήθειας σε αυτή τη χώρα. Και αν θέλουμε μακροπρόθεσμα να επιλύσουμε όχι όλα τα προβλήματα του Αφγανιστάν, ε, αλλά να φτάσουμε σε κάποια αξιοπρεπή κατάσταση όσον αφορά τη βοήθεια στη χώρα αυτή, να υπάρξει κάποια ρύθμιση των προβλημάτων της χώρας, ώστε το Αφγανιστάν να φτάσει στο επίπεδο των άλλων, πολλών άλλων φτωχών χωρών της χώρας, γιατί τώρα είναι κάτω από τις άλλες φτωχές χώρες του κόσμου. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν από εδώ, από τις δυνατότητες που έχουμε εμείς να αλλάξουμε το Αφγανιστάν στο μέλλον και η δική μας δυνατότητα είναι η βοήθεια την οποία παρέχουμε στο Αφγανιστάν. Και ε, με την έκθεσή μου και τις προτάσεις ε, που κάνουμε, ακριβώς αυτό θέλουμε να επιτύχουμε. Για την ειρηνευτική διαδικασία, η πρότασή μου είναι να υποστηρίξουμε πλήρως την ειρηνευτική διαδικασία, διότι είναι η μόνη εναλλακτική λύση στον πόλεμο του Αφγανιστάν. Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν ε, βρίσκεται σε μια στάσιμη κατάσταση. Δεν υπάρχει, κανείς δεν έχει προοπτική τελικής νίκης σε αυτή τη σύραξη. Οι Ταλιμπάν δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσουν γιατί οι διεθνείς δυνάμεις μπορεί να παραμείνουν στο Αφγανιστάν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι διεθνείς δυνάμεις επίσης ποτέ δεν θα κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο, γιατί είναι αδύνατο ε, να διεξαχθεί ένας ε, τέτοιος ασύμετρος πόλεμος σε αυτή τη χώρα. Και αυτή είναι και η γνώμη των ίδιων των στρατιωτικών. Μιλήσαμε με τους επικεφαλείς, με το, στρατηγό, ε, με το επιτελείο του στρατηγού Μακρίσταλ και γνωρίζουν ότι πρέπει να υποστηρίξουν την ειρηνευτική διαδικασία και ότι πρέπει να έχουν τη συνένεση του λαού του Αφγανιστάν. Και η ειρηνευτική διαδικασία σημαίνει ότι χρειάζεται μια νέα κυβέρνηση εθνικής ενότητας που μπορεί να προκύψει από ως αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ της κυβέρνησης Καζάη και των Ταλιμπάν από την πλευρά των ε, Ευρωπαίων ε, τονίζω ότι υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις για μας, για να υποστηρίξουμε εμείς αυτή τη διαδικασία. Πρώτον, ε, η απαγόρευση της, Αλκα... της δράσης της στην χώρα. Δεύτερον, πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του συντάγματος του Αφγανιστάν. Και τρίτο σημείο, ε, η ε, πάυση καλλιέργειας οπιούχων που είναι η πιο σημαντική ε, ζημιά που κάνει το Αφγανιστάν στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία θέτουμε ως προϋποθέσεις για συνομιλίες με τους συνομιλητές μας. Όσον αφορά την παρέμβαση στην αυτονομία της χώρας, δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντος, διότι στο παρελθόν προσπαθήσαμε να υπαγορεύσουμε τις ε, κινήσεις ε, της πολιτικής ακόμη και στο παραμικρό επίπεδο. Όσον αφορά την εκπαίδευση της αστυνομίας, η κατάσταση είναι πολύ κακή, υπάρχει μεγάλη σπατάλη. Τα τεράστια ποσά τα οποία έχουν μπει στον προπολογισμό για την εκπαίδευση της αστυνομίας ε, σπαταλήθηκαν και μέχρι πριν από ένα χρόνο στην Αμερικανική κυβέρνηση κανείς δεν ήξερε πώς δαπανήθηκαν 6 δισεκατομμύρια δολάρια για την εκπαίδευση της αφγανικής αστυνομίας, κανείς δεν ξέρει πού κατέληξαν. Γίνονται έρευνες στο Κογκρέσο για να βρουν ε, ε, ε, κάποια αίτια, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ανατίθεται σε ιδιωτικές εταιρείες η εκπαίδευση της αστυνομίας είναι ένα αίτιο. Πολλές από αυτές τις εταιρείες έχουν κακή φήμη. Υπάρχει η πρώην Blackwater και άλλες τεράστιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που έχουν, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ κακή φήμη και στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και τα περισσότερα προβλήματα δημιουργούνται ε, από την κακή εκπαίδευση που παρέχουν στην αφγανική αστυνομία. Υπάρχει και η ευρωπαϊκή προσέγγιση, δηλαδή το να στέλνουμε αποστολές όπως η eu στο Αφγανιστάν και υπάρχουν και μικρές εθνικές αποστολές στο Αφγανιστάν που εκπαιδεύουν ε, μικρό αριθμό Αφγανών αστυνομικών. Η πρότασή μου στην έκθεση υπάρχει και η αποστολή εκπαίδευση του ΝΑΤΟ που κατά τη γνώμη μου είναι η καλύτερη δομή που υπάρχει στο Αφγανιστάν για την εκπαίδευση της τοπικής ε, αστυνομίας και πρέπει να αποτελέσει το κέντρο μιας μελλοντική προσπάθειας για πραγματική εκπαίδευση της αστυνομίας. Σήμερα είναι απόλυτα μη ικανοποιητική αυτή η εκπαίδευση. Το 90% των Αφγανών αστυνομικών είναι αγράμματοι. ενώ το ποσοστό εγγραμματισμού της χώρας είναι 70%. Άρα, αφού είναι 70% οι υπόλοιποι αγράμματοι και 90% οι αστυνομικοί, είναι από το χειρότερο κομμάτι του πληθυσμού. Επίσης υπάρχει ε, μεγάλο μέρος ε, τοξικομανών και μετά την εκπαίδευσή τους, ε, πολλοί από τους αστυνομικούς φεύγουν και πηγαίνουν σε κάποιες άλλες πιεσίες ή εξαφανίζονται. Μας ενδιαφέρει λοιπόν ε, η εκπαίδευση των αστυνομικών και εγώ προτείνω μια ενοποίηση της εκπαίδευσης των αστυνομικών ε, στο πλαίσιο της δομής ε, του ΝΑΤΟ ούτως ώστε μέσα σε 2 τρία, τέσσερα χρονια να μπορέσουν τα ξένα στρατεύματα να αποχωρήσουν και να αφήσουν τους Αφγανούς με κάποιο ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας το οποίο θα μπορούν ήδη να παρέχουν στη χώρα τους. Για το θέμα της καλλιέργειας της παπαρούνας, που όπως σας είπα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας στην Ευρώπη, πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με τη Ρωσία, που λόγω του Αφγανιστάν έγινε η δεύτερη παγκόσμια αγορά οποίου από το Αφγανιστάν. Η πρώτη είναι η Ευρώπη με 1,5 εκατομμύριο ε, τοξικομανείς ε, και στη Ρωσία είναι 2 εκατομμύρια οι τοξικομανείς, που είναι διπλάσιο το ποσοστό από στην Ευρώπη δεδομένου του πληθυσμού της Ρωσίας. Οι Ρώσοι καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι η πηγή του προβλήματος του εθισμού και της τοξικομανίας είναι το Αφγανιστάν. Έχει δεκαπλασιαστεί το ποσοστό των τοξικομανών στη Ρωσία τα τελευταία δέκα χρόνια και θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια συμφωνία με τη Ρωσία γιατί τα βασικά θύματα του Αφγανιστάν είναι η Ευρώπη και η Ρωσία. Ενώ η Αμερική παίρνει την ηρωίνη της, προμηθεύεται την ηρωίνη της από άλλα μέρη του κόσμου. Είναι απόλυτα απαραίτητη λοιπόν μια συμφωνία με τη Ρωσία και θα πρέπει να καταρτήσουμε ένα σχέδιο για την εξάλληψη της καλλιέργειας της παπαρούνας. Ε, έχω μιλήσει και με τους υπεύθυνου της αναπτυξιακής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών και νομίζω ότι ε, μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Το πρόβλημα είναι η παραπληροφόρηση, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι πριν από 20 χρόνια η καλλιέργεια παπαρούνας ε, κάλυπτε όλη την Ασία και σιγά σιγά ξεριζώθηκε από παντού εκτός από το Αφγανιστάν. Έχει καταργηθεί στην Τουρκία, έχει καταργηθεί στο Πακιστάν ε, που προηγήθηκε του Αφγανιστάν ως κύριος προμηθευτής ε, παγκοσμίω. Έχει εξαλειφθεί στο Λάος όταν ήμουν εγώ υπεύθυνο σε αυτήν την υπηρεσία και στο Βιετνάμ και στην Ταϊλάνδη. Το πρόβλημα τώρα λοιπόν είναι το Αφγανιστάν είναι ο πιο σημαντικός προμηθευτής ε, μήκονος της υπνοφόρου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το, μπορούμε να ε, διαθέσουμε το 10% των ποσών που διαθέτουμε παγκοσμίω για το Αφγανιστάν και αυτό είναι ένα ποσό που θα αρκέσει ε, για την εκρίζωση του προβλήματος των οπιούχων. Αν θεσπίσουμε ένα τέτοιο μέτρο, είμαι πεπισμένο ότι μπορούμε να δούμε κάποιο φω στην κρίση του Αφγανιστάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αλλά όταν αναφέρεστε χώρες όπως η Ταϊλάνδη και άλλες που πέτυχαν, καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν αρχές εκεί, ε, μηχανισμοί, ε, θεσμοί που χρειάστηκαν υποστήριξη μεν, αλλά στο Αφγανιστάν ακόμα είναι προσίδρυση αυτή ε, αυτοί οι θεσμοί και οι οργανισμοί και οι μηχανισμοί. Δεν υπάρχουν καν. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε είναι ευπρόσδεκτο. Αλλιώς το πρόβλημα θα παραμείνει. Τώρα, η κυρία Νικόλ Κιλ ζήτησε το λόγο διότι πρέπει να πάει ε, σε άλλη συνεδρίαση και θα ε, δεχτώ να μιλήσει. Ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη. Πρέπει να φύγω να πάω να ψηφίσω σε άλλη επιτροπή. Θα ήθελα όμως να πω στον κύριο Αρλάκη ότι η προσέγγιση του για το Αφγανιστάν και τη διεθνή παρουσία δεν είναι καθόλου συγκαταβατική ήταν και σας ευχαριστώ γι' αυτό πάρα πολύ ειλικρινής ο απολογισμός σας για την παρουσία μας στο Αφγανιστάν, τη στρατηγική, την οικονομία, τη συνέπειες, την παγίδα αυτή που μας ε, έριξε η πολιτική ε, του Προέδρου Μπούς. Τώρα, το ερώτημα είναι τι να κάνουμε για να αποχωρήσουμε το συνομότερο. Γιατί ε, σύμπασα η κοινή γνώμη διεθνώς επιθυμεί να φύγουμε. Όλοι οι πολίτε ζητούν να γυρίσουν πίσω τα στρατεύματα και στην Ευρώπη και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Τι να κάνουμε λοιπόν για να βγούμε από την παγίδα αυτή το συντομότερο δυνατό, χωρίς βέβαια να εγκαταλείψουμε τους Αφγανούς ε, στη μοίρα τους. Να επανέλθει η χώρα στην κατάσταση που ήταν πριν από 10 χρόνια. Τι να κάνουμε λοιπόν έτσι έστω η τόσο σημαντική οικονομική επένδυση την οποία επισημάνατε για αυτές οι ανθρώπινες απώλειες που είναι πάρα πολλές, υπερβολικά πολλές και ε, στους Αφγανούς και ε, ε, στους δικούς μας στρατιώτες να μην είναι μια τρύπα στο νερό. Πώς θα φύγουμε από το Αφγανιστάν χωρίς να παραδώσουμε τη χώρα στους Ταλιμπάν και στην πρώτερη κατάσταση. Είναι γεγονός ότι έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα λάθη από τους Αμερικανούς. Εμπιστεύτηκαν υπερβολικά τον κύριο Καρζάη που δυστυχώς δεν ήταν πάρα πολύ αξιόπιστος ο άνθρωπος. Το έλεγαν κάποια από το παρελθόν. Ε, υπάρχει διαφθορά στην ίδια την κυβέρνηση της χώρας. Ο Καρζάη θεωρείται ότι έχει κάνει νοθεία στις εκλογές ε, η κυβέρνηση δεν έχει κύρος. Είναι πραγματικά ένα πρόβλημα η αδυναμία της κυβέρνησης. Οι Αφγανοί δηλώνουν ότι χρειάζονται ακόμα τη διεθνή παρουσία ως προστασία και χέγγιο για να τον παρακαλουθούν και να μην τον αφήνουν το καρσάι να κάνει ό,τι θέλει. Και ό,τι να είναι και υπερβολικές παραχωρήσεις προς τους Ταλιμπάν. Γνωρίζουμε και το ρόλο του Πακιστάν στη σύγκρουση αυτή και θα πρέπει να φεθεί ε, να επιβάλλει τη γνώμη του μόνο του. Και πάλι αντιμετωπίζουμε το θέμα των μειονοτήτων. Ο Καρσά είναι παστούν και ε, απομονώθηκε τελείως, δεν έλαβε υπόψη του ούτε τους Τατζίκους, ούτε τους Ουσμπέκους, ούτε τους Σαζαρά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και αυτό το ζήτημα του σεβασμού των μειονοτήτων και η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή έχω πει και στο παρελθόν ότι ένα από τα θέματα που έχουν σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η στήριξη σημαντικών προσώπων στο Αφγανιστάν, που δεν είναι ο κύριος Καρζάη βέβαια. Η κυρία Σορομπή, που είναι περιφερειάρχης του Μπαμιάν, και το λέω γιατί τη γνωρίζω προσωπικά. Την έχω γνωρίσει, είναι καταπληκτική γυναίκα, κάνει θαυμάσια πράγματα, πάρα πολύ θετικά είναι ε, ε, αζαρά ε, στην εθνότητα και δεν επενδύουμε αρκετά στην επαρχία, στην περιφέρεια. Δεν θα πρέπει όλα τα αυτά να πηγαίνουν στη σύγκρουση με τους Ταλιμπάν και στις περιφέρειες που είμαστε είναι γνωστές λόγω των εχθροπραξιών. Θα πρέπει να ενισχύουμε και τους περιφερειακούς ηγέτες όπως είναι η κυρία Σορόμπη, πολύ πιο θετικό και θα δώσει και ελπίδα στους Αφγανούς και θα τους δώσει ίσως και κέφι και όρεξη να κάνουν κάτι άλλο από το να καλλιεργούν την υπνοφόρο. Τώρα εγώ δεν θα τολμήσω να προβλέψω κάποια στρατηγική. Δεν θεωρώ καθόλου τον εαυτό μου ειδικό στις στρατιωτικές στρατηγικές. Προτιμώ την επικοδομητική πολιτική προσέγγιση. Ευχαριστώ τον εισηγητή ε, που θα συμπεριλάβει μερικά θέματα πρότεινα και εγώ για το ρόλο των γυναικών. Είναι αδιανόητο να εγκαταλείψουμε το Αφγανιστάν και να παραδώσουμε τις γυναίκες στους Ταλιμπάν. Θα πρέπει να επαγρυπνεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις γυναίκες στα δικαιώματά τους που δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Έχει γίνει λοιπόν πρόοδος. Θα δούμε τι θα γίνει στη διάσκεψη ε, που επίκειται στην Καμπούλ σε λίγες μέρες. Μάθαμε ότι διακόπτει προσωρινά τη βοήθεια Ευρωπαϊκή Ένωση στα 600 εκατομμύρια για να πιέσει την κυβέρνηση Καρζάη και να δεσμευτεί και να δώσει και σημεία ε, γραφής ότι καταπολεμά τη διαφθορά, τη ότι γίνονται πρόοδοι στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα γυναικεία δικαιώματα. Δεν μπορούμε να θυσιάσουμε τις γυναίκες ε, για να γίνει ειρήνη με τους Ταλιμπάν ή τους πρώην Μουτζαχεντίν και τους πολέμαρχους. Αυτά. Τα ξέρει ο κύριος Αρλάκη, ε, κατά τα άλλα πάρα πολύ θετική, ειλικρινή, σε παραλαμβάνω, ε, ε, ικανοποιητική. Δεν διστάσατε να ομολογήσετε και τις αποτυχίες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα παρακαλέσω τους επόμενους ομιλητές να συντομεύσουν κάπως με τις παρατηρήσεις τους. Ο κύριος Μπρέντα λοιπόν, που αντικαθιστά τον κύριο Κασουλίδη σκιώδη ηγητή για το ΕΛΚ. Κύριε Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αντικαθιστώ τον κύριο Κασουλίδη που είναι υπεύθυνο για την ε, αποστολή αυτή ο Σκιώδης από την πλευρά της δικής μας ομάδας και θα ευχαριστήσω εδώ τον εισηγητή για την εξαιρετική του έκθεση και τις παρατηρήσεις που μας επέβαλε. Τώρα έχω και εγώ κάποιες ε, δικές μου, δικά μου σχόλια για την έκθεση αυτή. Κάποιες Σίγουρα θα χρειαστεί να υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες, όμως έχουμε αρκετό χρόνο γι' αυτό ούτω ή άλλω, μέχρι τον Σεπτέμβριο. Οπότε η πρώτη μου παρατήρηση αφορά τον τίτλο Νομίζω καλό θα ήταν να παραμείνουμε στον αρχικό τίτλο, δηλαδή μια νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Αφγανιστάν. Εάν διαγραφεί ο όρος Ευρωπαϊκή Ένωση, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρωπαϊκή προοπτική χάνεται. Κάτι που δεν με βρίσκει σύμφωνο, θα πρέπει να δοθεί έμφαση εκεί Οπότε καλό θα ήταν να συμπεριληφθεί ξανά ο όρος EU Strategy, στρατηγική της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τίτλο ήδη. Δεύτερη παρατήρηση. Παρατήρησα ότι το πρόγραμμα δράσης του Συμβουλίου για το Αφγανιστάν αναφέρεται στην αρχική εκδοχή μεν, αλλά δεν τονίζεται αρκετά στη συνέχεια της έκθεσης. Νομίζω ότι το στοιχείο αυτό θα πρέπει να εμφανίζεται με μεγαλύτερη έμφαση και στο υπόλοιπο κείμενο, γιατί είναι καθοριστική σημασία. Εδώ υπάρχει επίσης ένα παράθεμα του Καρλ Μπίλτ, μια δήλωση η οποία είναι σημαντική, προέρχεται από το 2009, είναι και πολύ χρήσιμη για το γενικότερο αρχιτεκτόνημα, τη διάρθρωση του κειμένου. Κατά τρίτον, διαπιστώνω ότι θα πρέπει να δούμε και το ιστορικό πλαίσιο της σημερινή κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στο Αφγανιστάν και βρίσκω ότι η έκθεση είναι πολύ ευγενική, πολύ γενναιόδορη με τους Ταλιμπάν. Στη σελίδα 37 λέγεται ότι οι Ταλιμπάν κατάφεραν να εξαλείψουν, να καταπολεμήσουν την κουλτούρα του, της καλλιέργειας οποίου. Εδώ στην παράγραφο 30. 5 λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει η διατύπωση. Και το ίδιο και στην παράγραφο 59 για την κυβέρνηση Μπούς και τα προβλήματα τα σχετικά με την καλλιέργεια οποίου. Η κυβέρνηση Μπούς ούτως ή έχει παρέλθει. Είναι περασμένα ξεχασμένα αυτά Θα έπρεπε λοιπόν να αφιερώσουμε μια παράγραφο ολόκληρη για να μιλήσουμε για δεδομένα που σήμερα συναντώνται επί τόπου. Μια ολόκληρη παράγραφο για να επικρίνουμε την κυβέρνηση Μπούς δεν μου φαίνεται απαραίτητη. Και ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα προς τον εισηγητή. Ποιες είναι οι πηγές στις οποίες στηρίζεται τα λεγόμενα των παραγράφων 12 και 13 αναφέροντας τις παραγράφους αυτές ότι πέντε ημέρες πολέμου ως προς το κόστος θα έφταναν για να εξαλείψουμε την φτώχεια. Και ότι θα μπορούσαν να χτιστούν 6.000 σχολεία εάν χρησιμοποιούσαμε τα σπόρους για να δοτηθεί μια εβδομάδα πολέμου. Ποια είναι η εξοπιστία των υπολογισμών αυτών, πού βρήκατε τα αριθμητικά στοιχεία και τι σχέση έχουν με το υπόλοιπο κείμενο. Δεν νομίζω ότι αρκεί να έχει κανεί πολλά κονδύλια στα χέρια του για να τα καταφέρει όλα αυτά και να τα επιτύχει. Είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα και το ξέρουμε όλοι. Γιατί λοιπόν αυτέ οι τόσο εύκολε αναφορέ. Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά το νόημα. Σχεδόν ολοκλήρωσα την παρέμβασή μου και νομίζω ότι στόχο θα πρέπει να έχουμε να καταλήξουμε σε μια ισόρροπη έκθεση που να παρουσιάζει σωστά την ευρωπαϊκή πολιτική ως προς το Αφγανιστάν. Αυτή θα πρέπει να είναι η γραμμή που θα μας οδηγήσει στην σύνταξη της έκθεσης αυτής για το Αφγανιστάν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Νόιζερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η έκθεση του εισηγητού μας πίνω αρλάκι, δείχνει ότι έχει προετοιμάσει το κείμενό του με πολύ μεγάλη ικανότητα, πολύ μεγάλη εμπειρία και πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και συμπεριέλαβε και τις δικές μας προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Η πολιτική κατεύθυνση ε, της έκθεσης σε γενικές γραμμές είναι σωστή, Τέσσερις είναι άξονες, διεθνής βοήθεια, ειρηνευτική διαδικασία, εκπαίδευση της αστυνομίας και καταπολέμηση της καλλιέργειας ε, της ε, Παπαρούνας. Για τη διεθνή βοήθεια νομίζω είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα και πάρα πολύ πενιχρά τα αποτελέσματα σχεδόν καμία βελτίωση δεν έχει επέλθει στη καταπολέμηση της φτώχειας, στη ε, βρεφική ή μητρική θνησιμότητα. Και επίσης είναι και μια έκθεση που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα ε, ή μάλλον την αναποτελεσματικότητα της διεθνούς οικονομικής βοήθειας. Και χαίρομαι που αυτό το εξηγεί στη παράγραφο 12 και 13. Δηλαδή πόσα χρήματα κατασπαταλώνται και πάνε χαμένα, ενώ θα μπορούσαν να είχαν πιάσει τόπο. Το δεύτερο κεφάλαιο, η νευτική διαδικασία. Θα πρέπει να πούμε ότι ο βασικός στόχος επετεύθη να εκδιωχθεί η Αλκάιντα, που ήταν όντως ο πρώτος στόχος. Και επόμενη στόχη είναι η επιβολή του συντάγματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά βλέπουμε να επανέρχεται η καλλιέργεια της υπνοφόρου Μύκονος. Στην εκπαίδευση αστυνομία θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν επιτύχαμε το στόχο μας Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Εδώ και χρόνια δεν καλύπτουμε τους στόχους ε, που έχει θέσει η UPOL, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική ε, Δύναμη εκεί. Και θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι αποτύχαμε. Εγώ θα ήθελα εδώ να έχουμε και γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης για την αναπτυξιακή βοήθεια, όπου είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει σαφής διαχωρισμός οπωσδήποτε της ε, στρατιωτικής βοήθειας με την πολιτική βοήθεια. Ε, ότι ακόμα και όταν θα έχουν αποχωρήσει τα στρατεύματα, θα πρέπει να συνεχίζεται και η πολιτική βοήθεια, που δινόταν έτσι κι αλλιώς και πριν το 2001. Και μετά το 2014 θα χρειαστεί να συνεχιστεί ενίσχυση, πολιτική όχι στρατιωτική επαναλαμβάνω. Και πολλές ε, οργανώσεις βοηθείας μου είπαν ότι και για λόγους ασφαλείας ε, χρειάζονται σαφή διαγορισμό ποια βοήθεια πηγαίνει σε στρατιωτικούς σκοπούς και ποια σε πολιτικούς. Ένα πρόγραμμα, πρόβλημα συγγνώμη, βασικό που έχουμε και παραμένει είναι η καταπολέμηση ε, της διαφθοράς. Αν θεωρούμε ανεξάρτητη χώρα το Αφγανιστάν, θα πρέπει να διαχειρίζονται τη βοήθεια αυτή η ίδια Αφγανή ή τουλάχιστον ένα τμήμα της, αλλά με πολύ σημαντικούς ε, μηχανισμούς ελέγχου για να καταπολεμάται και να περιορίζεται η διαφθορά. Στην ευτική διαδικασία συμφωνούμε απολύτως ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και κάποιο τρόπο του Ταλιμπάν, αλλά να κάνουμε μια διάκριση. Τι είναι η Ταλιμπάν, 7, 8, 10 διαφορετικοί πολιτικοί σχηματισμοί. Είναι οι σκληροπυρηνικοί, οι ακεραιόφρονες μέχρι και ε, πρόσωπα της κοινωνίας των πολιτών που στις περιφέρειές τους δεν έχουν ε, άλλη δυνατότητα παρά να συνεργάζονται με τους Ταλιμπάν ή να εξαγοράζονται από τους Ταλιμπάν. Ε, ένα πρώτο τελευταίο σχόλιο. Στις αστυνομικές αποστολές έχω πολύ μεγάλες επιφυλάξεις ως προς την πρόταση αυτή να μπει υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ η αστυνομική δύναμη. Όχι. Και εδώ χρειάζεται σαφής διαχωρισμός, άλλη αποστολή του ΝΑΤΟ και άλλη αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση ενός κράτους δικαίου και σε ό,τι αφορά την περιφερειακή διάσταση θα πρέπει περισσότερο να συμπεριληφθούν και το Πακιστάν και η Ρωσία αλλά και το Ιράν που είναι πολύ σημαντική γειτονική χώρα. Από δική μας πλευράς επαναλαμβάνω θα κάνουμε επιπλέον ε, τροπολογίες και προτάσεις πάντως σε γενικές γραμμές είναι σωστή η πολιτική κατεύθυνση της έκθεσης. Και ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή κύριο Αρλάχη. Ευχαριστούμε ο κύριος Μάγερ, ο Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Αρλάκη. Στην ομάδα μου αξιολογούμε θετικά την προσέγγιση της έκθεσης σε αυτό το λαβύρινθο του Αφγανιστάν που μας έχει βάλει ο πρόεδρος Μπούς και δεν βρίσκουμε ούτε λύση, αλλά δεν βλέπουμε και διέξοδο. Πολιτικά ο κύριος Ομπάμα στο Κάιρο διαχώρισε τη θέση του και έκανε μια μεγάλη δήλωση πολύ σημαντική ε, και είχε και μεγάλη ε, απήχηση στον αραβικό κόσμο ότι καμία χώρα δεν μπορεί να επιβάλλει το σύστημά της σε μια άλλη χώρα. Έγινε μεγάλη φασαρία μετά από 9 χρόνια. Δεν έχουμε πετύχει κανένα στόχο, κανένα στόχο όμως. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε διέξοδο και λύση οι ημερομηνίε είναι δεδομένε. Αρχίζει η παράδοση των εξουσιών ήδη από τον Ιούλιο του 2011 με αποχώρηση των πρώτων Αμερικανικών στρατευμάτων, αλλά ο κύριος Πετρέους, ε, ο νέος ε, διοικητής, ε, δήλωσε στο ΝΑΤΟ και στη Γερουσία ότι τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει ακόμα, είναι μπροστά μας. Ο Ιούλιος ήταν χείριστος μήνας για τα στρατεύματα, 102 ε, πεσόντες ε, στο πρώτο εξάμεινο 320 τα θύματα ήδη των στρατιωτών και επί χίλια ε, πολλαπλασιάζονται τα θύματα του αμάχου πληθυσμού, τα αθώα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Μιλήσατε για τις βοήθειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέβαλε μέχρι το Σεπτέμβριο, ανέστηλε την πληρωμή των 600 εκατομμύρων περιμένοντας τη διάσκεψη και η Γερουσία των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι από τα 2-3 δολάρια, 2, συγγνώμη, ε, ε, τα περισσότερα δίνονται για προστασία μαφιόζων και Ταλιμπάν. Αυτό το ομολογεί η ίδια η Γερουσία. Άλλο ένα στοιχείο σε αυτό το λαβύριθο. Έχουμε τη βοήθεια για την ανοικοδόμηση, αλλά ολόκληρα δισεκατομμύρια δεν φτάνουν ποτέ στην ανοικοδόμηση. Και κλείνει όλο και περισσότερο ο λαβύρινθος και απομακρύνεται ακόμα περισσότερο η έξοδος. Κύριε Αρλάκη, βεβαίω το είπατε κι εσείς ότι δεν είναι στρατιωτική η λύση, αυτό είναι σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Ο στρατηγός Πετρέος ε, δεσμεύτηκε να μειωθούν τα θύματα ε, μεταξύ των αμάχων, γιατί όσο περισσότερα είναι τα θύματα μεταξύ των αμάχων, αυξάνονται ε, οι αντάρτες. Γι' αυτό είναι παράλογο ε, να γίνονται αυτοί τυφλοί βομβαρδισμοί. όσο ακολουθούν αυτή την τακτική, τόσο θα αυξάνονται οι γραμμές των ανταρτών. Όταν βλέπει κάποιο να σκοτώνεται ολόκληρη η οικογένεια, να κατακρεουργείται από ένα βομβαρδισμό που προέρχεται από 10.000 μέτρα και πλέον, φυσικά θα πάει να ενταχθεί στου αντάρτε. Θα πρέπει να συμμετέχει η Ρωσία, η Κίνα και το Πακιστάν. Ε, ε, στην προσπάθεια αυτή να πούμε να σταματήσει η κατοχή η κυβέρνηση ε, δεν έχει δημοκρατική νομιμότητα και την έχει διαποτίσει η διαφθορά, δεν υπάρχουν σωστοί μηχανισμοί που να αποδεικνύουν ότι τα χρήματα πηγαίνουν στην εκρίζωση της φτώχειας, όλα αυτά που είπατε κύριε Σιγητά, ε, στην εκρίζωση ε, της καλλιέργειας οπιούχων και στην πραγματική ανοικοδόμηση μιας κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο η Ρωσία η Κίνα και το Πακιστάν και να λυθεί και επιπλέον και ε, η σύγκρουση στο Κασμίρ μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Το 2011 είναι αύριο, ε, σε ένα χρόνο. Ε, μας μένει ένας χρόνος να, να ψάξουμε την έξοδο από το τούνελ έτσι ώστε να αποχωρήσουν τα στρατεύματα και να εξαφανιστούν από το Αφγανιστάν η διεθνής κοινότητα να βοηθήσει την ανοικοδόμηση αλλά την ουσιαστική. Η ομάδα μου θα εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή, να βοηθήσει, να συνεργαστεί στην έκθεση που είναι στη σωστή κατεύθυνση, επαναλαμβάνω, για να δούμε αν μπορεί να συνεισφέρει με τριοπαθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βρούμε την έξοδο από το τούνελ, στο, στην οποία μας έσπρωξε δούνελ ο πρόεδρος Μπούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Yes. Um, Mr. please. Ευχαριστούμε κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, με την ε, συμφωνία σας. Θα ήθελα να πάρω το λόγο στους ηγητής της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και να προσεγγίσω το όλο θέμα από την οπτική γωνία των θεμάτων της δικής μας Επιτροπής και της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικώ. Κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Όταν μιλάει κανείς για το ζήτημα του Αφγανιστάν, τίνει να αναφέρεται και στο στρατηγό Ντεγκόλ που έλεγε ότι για να πάω στην Ανατολή που είναι τα πράγματα τόσο περίπλοκα έπρεπε να έχω το μυαλό μου ξεκάθαρο. Έτσι λοιπόν, όσο λίγο περισσότερο κοιτάει κανείς το Αφγανιστάν, τόσο αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα είναι σχετικά απλά εκεί. Η Καμπούλ, δεδομένων των συνθηκών, είναι μια πόλη που λειτουργεί λίγο πολύ ομαλά, ε, κάτι που δεν είναι απλό. Και αυτό το γνωρίζουν όσοι έχουν ε, μείνει στο Αφγανιστάν τα τελευταία χρόνια. Τώρα για τις γυναίκες που έχουν το θάρρο να φορέσουν και κραγιόν ή για ανθρώπους που πηγαίνουν στο θέατρο, για τις γυναίκες που βγάζουν την μπουρκα, καταλαβαίνετε ότι αυτή η πρόοδο είναι τεράστια. Δεν ξέρω αν αυτά μπορούν να καταμετρηθούν στατιστικώς, αλλά σίγουρα υπάρχει πρόοδο. Οι Αφγανοί, ιδίω οι γυναίκε τολμούν τολμούν να προβάλλουν την προσωπικότητά τους, κάτι που στο παρελθόν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Η εικόνα λοιπόν είναι γεμάτη αντιφάσεις. Ο κ. Καζάη το 2004, όταν τον συνάντησα ως υπουργό Αμήνης, μου είπε σε πέντε χρόνια δεν θα χρειαζόμαστε πλέον κανέναν. Η χώρα μας θα είναι αυτάρκης από άποψη παραγωγής τροφίμων, η διεθνής βοήθεια θα είναι πλέον περιττή και τώρα βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Ε, τουλάχιστον σε επίπεδο αφγανικής ηγεσία, σίγουρα υπήρξαν αρκετές, ε, αρκετά σφάλματα, δηλαδή δεν έπεσαν μέσα στις προσβλέψεις τους. Τώρα, η αρχή της ιδιοποίησης, τι καταφέρνουμε ουσιαστικά να οδηγήσουμε του Αφγανού να αναλάβουν μόνοι του τον εκδημοκρατισμό λόγω χάρη τη χώρας. Αρκεί κανείς να κοιτάξει τι έγινε με τις πρόσφατες εκλογές που φαίνεται περισσότερο νοιάζαν με φαρσοκομωδία. Ο Καρζάη ε, πήρε την εξουσία, αλλά όχι ο λαό ε, ο λαός δεν ανέλαβε την ευθύνη της δημοκρατικής διαδικασία Υπάρχει απόσταση των φωτό μεταξύ των δύο καταστάσεων. Επιπλέον, στο Αφγανιστάν δεν φαίνεται καμία σαφή προοπτική για να μπορεί κανεί να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Τώρα για την ανθρωπιστική κατάσταση, το είπε και ο κύριο Αρλάκη στην εισαγωγή του. Το πιο αξιόπιστο κριτήριο, που είναι και το πιο εύκολο για το τι συμβαίνει σε μια χώρα γενικότερα είναι το ποσοστό θνησιμότητα των νηπίων κατά των 5 ετών. Είχαμε 250 από το 2005 και το ποσοστό αυτό τίνει να αυξάνεται. Γιατί το κριτήριο αυτό είναι εύγλωτο, γιατί ακριβώ δείχνει τι γίνεται με την κατάσταση των γυναικών, με τι νοσοκομιακέ ε, υποδομέ για τον ε, αλφαβητισμό και εάν. Αυτό σημαίνει ότι ένα τέτοιο ποσοστό ε, δίνει το αποτέλεσμα το εξή. Αν γεννηθούν χίλια παιδιά το 2010, θα έχουν πεθάνει 250 το 2015. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν λοιπόν αρκετοί γιατροί, αρκετέ υποδομέ και αρκετή ανάπτυξη. Και παραμένω σε αυτό το κριτήριο και μόνο για να μην μακρηγορήσω. Σε ό,τι αφορά την ε, παραγωγή. Α μην είμαστε υποκριτέ εδώ. Εάν βρισκόμασταν ε, στο Αφγανιστάν, θα είχαμε και εμεί ε, πέσει θύματα τη διαφθορά. Περισσότερο και από του Αφγανού, ίσω στις 15 του μήνα, όταν κανεί δεν ξέρει πώς θα βγάλει το μήνα στο τέλο του, κάτι προσπαθεί να κάνει. Όπω έλεγε και ο Κολλή, ο Γάλλο Κομίκος, ε, οι πιο δύσκολε μέρε του μήνα είναι 8 τελευταίε. Οι 20 τελευταίε. Έτσι λοιπόν μιλάμε για διαφθορά της ε, επιβίωσης και για την ε, διαφθορά των αρπακτικών, αν θέλετε, των μεγάλων οργανωμένων εγκληματιών. Η διαφθορά της επιβίωσης είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, αν η οικονομία μιας χώρας ε, βασιζόταν στο δίκαιο, ε, όπως ε, συνέβαινε παλιότερα ίσως σε χώρες όπως το Ζαΐρ, όταν ε, η οικονομία τη χώρα βασιζόταν στην εξωτερική βοήθεια και συγκεντρώνονταν στα χέρια λίγων, τα πράγματα αυτά ήταν τελείω διαφορετικά. Όμω, ο κρατικό έλεγχο του Αφγανιστάν μπορεί να ασκηθεί σωστά όταν ο Καρζάη από την αρχή τη προεδρία του δεν ελέγχει παρά μόνο την πρωτεύουσα, την Καμπούλ. Μιλάμε εδώ για συνθήκε που ισχύουν μόνο και αποκλειστικά για την Καμπούλ. Αλλά όταν είναι έτσι κατάσταση για έναν αρχικό κράτο, τα πράγματα δείχνουν ότι πολύ πρόοδο απομένει να γίνει. Ε, και για την θετική κατάσταση που σχετίζεται μέσα με τα ανθρωπιστικά. Το πρόβλημα όσων εργάζονται στα ανθρωπιστικά είναι ότι δεν μπορούν να προβλέψουν τι θα συμβεί τα προσεχή χρόνια. Γνωρίζουν ότι την ημέρα που θα φύγουν τα στατεύματα θα χρειάζονται ακόμα την παρουσία τους παρόλα αυτά. Και εδώ για να συντομεύω θα πω ότι το μεγάλο πρόβλημα του Αφγανιστάν μπορεί να συνοψιστεί σε δύο φράσεις. Στο Αφγανιστάν έχουμε στρατεύματα και ανθρωπιστικούς εργαζομένους με στρατιωτική στολή, ένστολους και χωρίς ε, στολή. Οι πολίτες εκπροσωπούν μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή ιδρύματα που δεσμεύονται από τις αρχές του διεθνούς δικαίου των ανθρωπιστικών οργανώσεων γενικότερα. Όμω αν του εξομοιώνουμε με τη στρατιωτική δράση, τα πράγματα περιπλέκονται. Υπάρχουν μάλιστα ανθρωπιστικέ οργανώσει που αρνούνται, αρνούνται οποιαδήποτε στήριξη, οικονομική στήριξη από τα κράτη για να μην ε, πληγεί η στάση αμεροληψίας ουδετερότητας που θέλουν να τηρήσουν. Αντιθέτως, άλλοι κατά καιρούς χρειάζονται στρατιωτική προστασία δεν φοβούνται δηλαδή τόσο το συσχετισμό, όμω δεν μπορούμε να του εντάσσουμε όλου στην ίδια κατηγορία. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και σωστά το έχετε γράψει στο σχέδιο γνωμοδότησή σα, ότι πρέπει να περιορίσουμε την ανθρωπιστική δράση των στρατιωτικών, των στατευμάτων στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Αλλά σε κάποιε περιπτώσει, κανεί άλλο πέραν των στρατιωτικών δεν μπορεί να προσφέρει ε, ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτέ οι περιπτώσει όμω θα πρέπει να παραμείνουν εξαιρέσει, να είναι έκτακτε. Γιατί επί τόπου και επειδή τα πράγματα βρίσκονται πάντοτε στο χείλο τη εμπόλεμη σύραξη, οι εργαζόμενοι των ανθρωπιστικών οργανώσεων τη Γαλλία, λόγω χάρη, εξομοιώνονται με, τους, με τα γαλλικά στρατεύματα. Γιατί πολλέ φορέ ε, ασκούν για διπλή ιδιότητα οι δυνάμεις, οι εχθροί δηλαδή που βρίσκονται στο Αφγανιστάν ε, δεν κάνουν διάκριση μεταξύ φορτικών και ε, Γάλλων και Γάλλων που εργάζονται για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Ο κύριος Αρλάκη μίλησε και για τα ναρκωτικά. Πρόβλημα αδυναμίας να δώσουμε εναλλακτικέ λύσεις στον αγροτικό τομέα, διαβλέπω εδώ. Αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε βλέπουμε ότι οι διακινητές ηρωίνης χρησιμοποιούν ένα σύστημα επανάληψης κάποιων πρακτικών. Γίνονται αφοσιωμένοι έτσι οι γεωργοί, τους δίνουν ωφέλη τόσα ώστε να σκεφτούν αργότερα τον κίνδυνο. Οι γεωργοί δηλαδή παράγοντας ναρκωτικά δεν διακινδυνεύουν τόσο τη ζωή τους και επιβιώνουν έτσι που να μην είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν καλλιέργεια δεδομένου ότι η χώρα βρίσκεται και στα πρόθυρα του πολέμου. Ε, τώρα για τις αρχές της δράσης που προτείνεται, από αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας. Εδώ καλά να είχαμε αξιολόγηση πιο λεπτομερή, πιο εμπεριστατωμένη. Ακούω και πολλές διαφορετικές απόψεις. Και ξέρω ότι υπάρχουν ε, τεράστια κονδύλια που έχουν δαπανηθεί επί τόπου, αλλά έχουμε και πολλούς θανάτους πολιτών ε, μη ένστολων στην πράξη από τους εργαζομένους των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Και θα πρέπει μάλιστα να χαιρετήσουμε εδώ και την ηρωική ε, στάση των ανθρώπων αυτών. Τώρα, αν είναι αποτελεσματικέ οι δράσει μα, ε, σε κάποιε περιπτώσει είναι πολύ αποτελεσματικέ. Δεν θα πρέπει η αποτελεσματικότητα των μεν να διαλύεται και να μαυρώνεται από τη δράση κάποιων άλλων στο Αφγανιστάν. Τώρα για τα αποτελέσματα συμφωνώ μαζί σα, είμαι απογοητευμένο σε μακροοικονομικό τουλάχιστον επίπεδο για την οικονομία. Το Αφγανιστάν έχει τεράστιο φυσικό πλούτο και εάν δεν είχε ξεκινήσει αυτός ο φαύλο κύκλος τη διαφθοράς, τη ε, αρνητική διάθεση για επενδύσεις στο Αφγανιστάν, η χώρα αυτή θα είχε τα πάντα στα χέρια τη ε, για να πετύχει. Όσοι επισκέπτονται και για λίγο το Αφγανιστάν, γρήγορα διαπιστώνουν αυτό που είχαν διαπιστώσει και οι Σοβιετικοί στο παρελθόν. Και αυτό που διαπιστώνουν τώρα τα στρατεύματά μα. Ότι είναι άνθρωποι που έχουν ε, την επιθυμία να πετύχουν, αλλά δεν είναι. Ε, αλλά δεν τους βοηθάνε γιατί δεν τους ε, είναι ανεπιθύμητοι οι ίδιοι. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι εδώ προσπαθούμε να βρούμε οποιοδήποτε πρόσχημα για να φύγουμε στο δυνατόν γρηγορότερα από το Αφγανιστάν. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθούμε, βλέποντα από το πρίσμα τη Επιτροπή Ανάπτυξη τα πράγματα, ότι για όσους βρίσκονται στη χώρα πρέπει τουλάχιστον μέχρι να φύγουμε να μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται εκεί αποτελεσματικά. Εδώ τώρα κάποιες προτάσεις Ω συνήθω ε, στο σχέδιο γνωμοδότηση, έχουμε δικαίωμα να κάνουμε αρχικά κάποιε προτάσει και μετά γίνονται κάποια μαγειρέματα για να καταλήξουμε σε τροπολογίε. Εδώ λοιπόν κάποιε αρχικέ σκέψει θα προσπαθήσω να τι συνοψίσω, προσπάθησα να τι συνοψίσω και τώρα μια τελευταία παρατήρηση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακριβώ στο Αφγανιστάν. Μπορούμε να κοιτάζουμε προ το παρελθόν, αλλά εσεί, ε, πρόεδρε, φίλε Πρόεδρε, που είσαστε Υπουργό Αμήνη το ίδιο διάστημα με εμένα. ξέρετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Όπω και εγώ, υπήρχε αρχικά διάκριση μεταξύ της, ε, της διαρκούς ελευθερίας της Enduring Freedom για να εκριζωθεί η Al-Qaeda, επιχείρηση που ολοκληρώθηκε με επιτυχία αλλά όταν αυτό ε, ενώθηκε, συνενώθηκε με την επιχείρηση ΙΖΑΦ, τότε άρχισαν τα προβλήματα. Δηλαδή η δύναμη προστασίας των ε, αμάχων και των πολιτών συνενώθηκε με τη δύναμη ε, της καταπολέμησης της Αλκάιντα. Και εκεί άρχισαν τα προβλήματα. Στο επίπεδο των στατευμάτων, λοιπόν, που γενικώ κάνουν εξαιρετικό έργο, που σκοπεύουν να προστατεύσουν τον πληθυσμό τελικά λόγω της εγχώνευσης αυτής των δύο δυνάμεων ε, δεν έχουν καταλήξει στο βέλτιστο αποτέλεσμα. Δεν θα έλεγα βέβαια ολοκληρωμένως ότι είμαι αισιόδοξο. Αποφασισμένο είμαι, αλλά όχι αισιόδοξο. Ευχαριστώ, Σάρλα. Ένα από τα πλεονεκτήματα του να μεγαλώνει κανείς ηλικία είναι ότι καταλαβαίνει ότι εκ των υστέρων βλέπει αν είχε δίκιο ή άδικο σε κάποιες εκτιμήσεις. Αλλά και στο παρελθόν είχαμε άλλες προσδοκίες. Θα παρακαλούσα τον κύριο Βάγκελ τώρα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο προηγουμένως αλλά δεν είχα φανταστεί ότι θα μπαίναμε σε τέτοιες λεπτομέρειες στην ουσία της συζήτησης, γιατί θα μπορούσα και εγώ να πω πολλά αυτή τη στιγμή. Η έκθεση είναι πάρα πολύ εμπεριστατωμένη, ε, στραμμένη προς το μέλλον, πολύ μεστή. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω κι εγώ σε ευχαριστίες προς τον εισηγητή. Είναι και προκλητική η έκθεση, είναι και αντιφατική, έχει πολλά στοιχεία για τα οποία πολλοί προσπαθούν ε, να μην συζητούν, να τα αποσιωπούν και να τα συγκαλύπτουν σε συγκεχημένες εικόνες που δίνουν από το Αφγανιστάν. Προσωπικά ε, θεωρώ πολύ σημαντικό το συμπέρασμα που λέγει ότι τα πράγματα στο Αφγανιστάν παρά ε, τις την πολιετή ε, και ακριβή παρουσία και δέσμευση ε, της διεθνούς κοινότητας, άλλων οργανισμών και μεμονωμένων προσώπων, η κατάσταση λέγω επιδεινώνεται συνεχώς, δεν βελτιώνεται καθόλου 9 χρόνια μετά. αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Άλλη διαπίστωση και άλλο συμπέρασμα. Η διεθνής κοινότητα συχνά επενδύει σε λάθος θέματα. Χάνονται χρήματα και για μας τους Ευρωπαίους θα ήταν επίσης πολύ καλό να καθίσουμε να σκεφτούμε τι κάνουμε και πώς. Είναι σωστά όλα αυτά που κάνει η Ευρώπη Θα πρέπει να σκεφτούμε και το πώς δαπανώνται οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν πηγαίνουν για καλό σκοπό. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ ε, σε μερικές προτάσεις και πρωτοβουλίες για τη συνέχεια που θα δοθεί στην έκθεση αυτή. Θεωρώ πολύ σημαντικό να κάνουμε ακρόαση και να ακούσουμε εκείνους που πήγαν στο Αφγανιστάν τα τελευταία χρόνια με τις πιο διαφορετικές ιδιότητες. Δηλαδή, να ακούσουμε εκείνου που εκπαίδευσαν αστυνομικούς ή ε, ανθρωπιστική ε, βοήθεια ή υπευθύνου διαφόρων έργων. Αυτές οι μαρτυρίες θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να έχουμε καλύτερη εικόνα της κατάστασης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύω είναι το θεσμικό εκείνο όργανο που προσφέρεται για να υπάρξει μια αντικειμενική ε, ματιά στην κατάσταση στο Αφγανιστάν. Επίσης θα πρότεινα κάπου στην έκθεση, δεν ξέρω σε ποιο σημείο, να αναφέρουμε λίγο τη σχέση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στο Αφγανιστάν με την κρίση στη Μέση Ανατολή και το ότι η σύραξη στη Μέση Ανατολή αποτελεί ε, πρόσφορο έδαφος για τη δημιουργία διεθνούς τρομοκρατίας. Και μάλιστα ε, η Αλκάιντα σήμερα ενισχύεται, έχω την εντύπωση, παρά αποδυναμώνεται. Μην θα πρέπει να το λησμονούμε και αυτό το στοιχείο τη σύραξη στη Μέση Ανατολή, ότι εκεί γεννήθηκε η Αλκάιντα, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, το Ανατολικό είναι πάρα πολύ οξύ και όχι μόνο ε, για την περιφέρεια εκεί με τη στενή έννοια, μεταφέρεται, μεταδίδεται στο Ιράκ, στο Ιράν, αύριο δεν ξέρω σε ποια άλλη χώρα. Ένα τελευταίο σημείο Είπαμε ότι είναι πολύ σωστή η προσέγγιση του Συγητού, ότι ε, εξετάζει ε, από τη σωστή σκοπιά την κατάσταση στο Αφγανιστάν και καλά ε, λέει ότι χρειάζεται περισσότερη περιφερειακή συνεργασία. Και, να συμμετέχουν και χώρες της περιοχής για να γίνει και πιο εύκολα δεκτή η διεθνής παρουσία από το λαό του Αφγανιστάν ειρηνευτικά στρατεύματα, ανθρωπιστική βοήθεια. Ακόμα και αυτοί θεωρούνται κατακτητές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε ο κύριος Μάουρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτησή μας με τις διαστάσεις που έχει πάρει δείχνει ότι και εμείς όλοι ενδιαφερόμαστε για την έκθεση αυτή. Ε, μόνο και μόνο γιατί καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό το θέατρο ειρήνης και πολέμου παίζεται ίσως το πεπρωμένο του υπόλοιπου κόσμου. Αυτός είναι και ο λόγος που είχατε τόσες παρεμβάσεις και φαίνεται σχεδόν να θέλουν να συντάξουν τελείως εκ νέου την έκθεση του κυρίου Αρλάκη. Έχουμε εδώ μια προδιάθεση να συνεισφέρουμε στο έργο του εισηγητή που ούτως ή άλλως αυτής εξ αρχής είναι πολύ διεκδοτική. Σε κάποια σημεία συμφωνώ, σε κάποια όχι, αλλά με μια σύντομη παρέμβαση ήθελα να εκφράσω δύο παρατηρήσει για δύο θέματα ουσία που αφορούν όχι τόσο πολύ την ανάλυση που έχετε κάνει, αλλά τις προτάσεις σας. Πρώτα απ' όλα για τις διεθνείς δυνάμεις. Ήδη στο Αφγανιστάν βρέθηκα με την Επιτροπή Προπολογισμών ε, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας και τα προβλήματα εκεί είναι πολύ σοβαρά. Απλώς να σημειώσω ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση σε αυτά που λέει ο συνάδελφος. Δηλαδή το να προβλέψουμε μηχανισμούς διανομής μέσω πολυμερών ε, συστηματών για να ενισχυθούν κατά προτεραιότητα η κυβέρνηση και τα θεσμικά όργανα του Αφγανιστάν, αυτό από μόνο του είναι αντιφατικό. Διότι σε ένα άλλο σημείο της έκθεσης αναλύεται το ποια ακριβώ είναι η συμπεριφορά της σημερινής κυβέρνησης που συμπίπτει με τη συμπεριφορά της προηγούμενης. Άρα ως προς αυτό καλό είναι ο εισηγητή, και αυτό το δούμε και με ενδεχόμενε τοπολογίε, να σκεφτεί κατά πόσο μπορεί να γίνει ένα συνδυασμό ε, Ένα σημείο που λόγω χάρη επεσήμαναν αρκετέ με κυβερνητικέ οργανώσει και ένα σημείο που πολλοί τίνουμε να παραβλέπουμε. Κάτι που σε πολλές περιπτώσεις έχει φανεί καλύτερο από τις άλλες προσπάθειες, δηλαδή την, το χτίσιμο νοσοκομείων, σχολείων, ε, δρόμων, να γίνουν συγκεκριμένε δράσεις στο, στη χώρα. Αυτό και με τη συνδρομή ίσω κάποιων στρατιωτικών δυνάμεων, μεταξύ των οποίων οι ευρωπαϊκές. Έτσι κι αλλιώς δαπάνες ήταν πολύ πιο ελεγχόμενες πολλές φορές για μας από ό,τι για άλλους τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν στις προτάσεις μας να επικεντρωθούμε στο πώς μπορούμε να έχουμε δράσεις χρήσιμες για τους πολίτες μέσω των στασιωτικών και για το πρόβλημα των ναρκωτικών. Το σχέδιο που προτείνει ο συνάδελφος Σαρλάκη σε προοπτική πενταετίας Δεν ξέρω κατά πόσο θα παραμείνει από το πλαίσιο, αλλά θέλω να καταλάβω το εξή. Υπάρχει λόγο για τον οποίο αξίζει τον κόπο να βρίσκεται. Μάλλον, αν υπάρχει λόγο για τον οποίο αξίζει να βρισκόμαστε στο Αφγανιστάν, είναι ακριβώ αυτό. Δηλαδή, η έλλειψη αστάθειας που προκαλείται από την κατάσταση στο Αφγανιστάν είναι κάτι που μπορεί να μας αφορά άμεσα όταν βγαίνουμε από τα σπίτια μας και κυκλοφορούμε στον δρόμο, αλλά το ίδιο και με την κατανάλωση της ε, ηρωίνης και ναρκωτικών. Πολλά σχετίζονται με τα όσα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε με περαιτέρω τροπολογίε να ενισχύσουμε την κατεύθυνση που παίρνει η νομοδότηση, η οποία κατά τα άλλα είναι σωστή ούτως ή Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάλερ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Αρλάκη για το έγγραφό του, για, την, το σχέδιο έκθεση. Νομίζω ότι τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει και η ανάλυση που κάνει είναι πολύ σωστή. Ένα σημείο κλειδί είναι το ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε εφόσον έχουμε κάνει μια αρχική σωστή ανάλυση της όλης κατάστασης. Εγώ θα ήθελα μια συγκεκριμένη πρόταση να κάνω. Νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι ένα θέμα που είναι η καταλληλότερη ευκαιρία για να συνεργαστούμε με το Αμερικανικό Κογκρέσο και τη Μόσχα. Δηλαδή, εφόσον έχετε συντάξει ένα τόσο καλό έγγραφο, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή ώστε να συζητήσετε και με τους ε, ομολόγους μας στις ΗΠΑ και στη Ρωσία. Νομίζω ότι στο Κογκρέσο αυξάνεται η έλλειψη ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της επιχείρησης στο Αφγανιστάν. Ω προ το θέμα αυτό, ο πρόεδρος Ομπάμα έχει ήδη πέσει στην ε, παγίδα που είχε στήσει ο προκατοχός του. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον από κοινού μπορούμε να εξεύρουμε ε, ευφυείς εναλλακτικέ λύσεις στην απόσυρση μεταδεύματων από το Αφγανιστάν. Yes. Thank you. The problem is... Ευχαριστώ πολύ. Το πρόβλημα είναι ότι ε, αρχίζει η απόσυρση, προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη δημιουργία του κράτους και θα πρέπει κάποιος ε, να αναλάβει την ασφάλεια ή κάποιος να δηλώσει νικητής και να αποχωρήσει. Θα δούμε, θα δούμε. Κυρία Κόπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον συνάδελφο κύριο Αρλάκη για ένα έντιμο ε, και πολύ καθαρό κείμενο σχετικά με ένα θέμα που μας αφορά όλους όπως είναι το Αφγανιστάν. Ε, το Αφγανιστάν είναι το μεγάλο στίχημα για τις Ηνωμένε Πολιτείε του Προέδρου Ομπάμα αλλά και για την Ευρώπη. Ε, για τον Πρόεδρο Ομπάμα το στίχημα είναι να κερδίσει αυτό τον πόλεμο, ήταν από τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή παρόλο που ε, αναγγέλλονται αποχωρήσεις στρατιωτών, όχι μόνο από τι ΗΠΑ αλλά και από Ευρωπαϊκέ χώρε, από άλλε χώρε του ΝΑΤΟ, ε, η νίκη δεν φαίνεται ορατή, δεν φαίνεται πιθανή. Η εσωτερική κατάσταση παραμένει επίσης πάρα πολύ προβληματική. Η διεθνή κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε με μισή καρδιά τον πρόεδρο Καρζάη, μετά από εκλογές νοθείας, που όλοι αναγνωρίσαμε ότι ήταν τέτοιες, ε, θεωρώντας ότι είναι ο μόνος συνομιλητής που μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα. Όμως η διαφθορά, η απουσία κράτους δικαίου, η καταπίεση των μειονοτήτων, η δραματική θέση των γυναικών είναι κεντρικά προβλήματα που η διακυβέρνηση Καρζάη δεν μπορεί ή δεν θέλει να αντιμετωπίσει. Το βασικό όμως πρόβλημα, όπως διατυπώνει και ο συνάδελφος κύριος Σαρλάκη στην έκθεσή του, είναι η φτώχεια παρά τα τεράστια ποσά που έχουν δαπανηθεί στη χώρα αυτή. Το Αφγανιστάν έχει γίνει γενικά για τη διεθνή κοινότητα, ειδικότερα για την Ευρώπη, μία μαύρη τρύπα. Τόσο σε στρατιωτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο οικοδόμησης κράτους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο, όπως ορθά επισημαίνει η έκθεση, απαιτεί μια νέα στρατηγική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν επιπλέον λόγο με την παρουσία της UPOL, της ε, επιχείρησης ε, αστυνομίας, να τοποθετηθεί και να διατυπώσει σήμερα μια νέα στρατηγική που δεν αφορά μόνο την ασφάλεια, αλλά θα είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση για το μέλλον του Αφγανιστάν. Εκτός όμως από αυτή τη νέα στρατηγική που σωστά επισημαίνεται όπως είπα στο κείμενο, για την έξοδο αυτής της χώρας από την κρίση και από τη φτώχεια, χρειάζεται και ένα πολύ πιο καθαρό μήνυμα, κατά τη δική μου γνώμη, από αυτό που δίνει ο εισηγητής στον πρόεδρο Καρζάη. Τα προβλήματα είναι πολλά, οι ευθύνε τη διεθνού κοινότητα, κυβερνήσεων, μη κυβερνητικών οργανισμών είναι πολλά. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να χαϊδεύουμε αυτόν ο οποίο έχει αυτή τη στιγμή την ευθύνη τη χώρα, όπω είναι ο πρόεδρο Καρζάη. Ε, δεν μπορεί να απαλλαχτεί αυτή από την ευθύνη επειδή η χώρα βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Έχουμε λοιπόν, για να τελειώσω, γιατί η συζήτηση είναι πολύ μακρά, ε, ένα κείμενο που αποτελεί μια εξαιρετική βάση συζήτηση για μας. Έχουμε αρκετό χρόνο όλοι να έρθουμε με σημαντικές ε, τροπολογίες, ώστε να μπορέσουμε να στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα προς τους συμμάχους μας, αλλά και προς το Αφγανιστάν και προς τον Πρόεδρό του, για τη δική μας αποφασιστικότητα να τοποθετηθούμε πια καθαρά και χωρίς συμβιβασμούς στο θέμα του Αφγανιστάν. Ευχαριστώ. <clears throat> Mr. please. Ευχαριστώ. Κύριος Κατσίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Αρλάκη για την έκθεση αυτή. Και θέλω να τον ευχαριστήσω και γιατί ανέλαβε τόσο μεγάλη δέσμευση και έχει καταβάλει τόση προσπάθεια με ουσιαστικό τρόπο. Δεν ακολουθεί μια συμβατική προσέγγιση, που, τη συνήθη προσέγγιση που ακολουθούν μέχρι τώρα τα θεσμικά όργανα έναντι του Αφγανιστάν. Μέχρι τώρα ε, φαίνεται ότι ε, υπάρχουν πολλά ελλείμματα ε, σε αυτό που έχουμε κάνει στην πράξη. Η έκθεση αυτή είναι μια ολοκληρωμένη έκθεση με περιστατωμένα στοιχεία μιλάει και για τις αιτίε ε, της κρίσης και υποδεικνύει και κάποιο, κάποιο οδό εξόδου προς ε, εξόδου από την κρίση. Και επανέρχομαι σε κάτι που πρότεινε και ο κύριος Στάλια σε σχέση με την Ρωσική Δούμα και το Αμερικανικό Κογκρέσο. Εγώ δεν ξέρω καμία χώρα της οποίας να βρίσκονται οι στρατιώτες στο Αφγανιστάν και να μην ανησυχούν οι πολίτες και τα κοινοβούλια της χώρας της. Νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο οι συντονιστές να συζητήσουν το αν θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να καλέσει μία συζήτηση για το Αφγανιστάν, στην οποία, να συγκαλέσει μια συζήτηση στην οποία θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων. Πιστεύω ότι πολλές χρήσιμες ιδέες θα μπορούσαν να προκύψουν από μια τέτοια συζήτηση. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι πριν από λίγους μήνες είχαμε κάνει μια ακρόαση Και είχαμε ακούσει πολλού ε, οι οποίοι είχαν πάει στο Αφγανιστάν. Είναι πολύπλοκα τα προβλήματα του Αφγανιστάν και γι' αυτό επιμένω ότι οι εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο Αφγανιστάν θα πρέπει να μα ενημερώνουν τακτικά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει τακτικά να οργανώνουμε τέτοιες ε, συζητήσεις. Δεν αρκεί μόνο να το συζητάμε εμείς εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ή στην Υποεπιτροπή ασφάλειας και άμυνας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητείτε ε, και στην Επιτροπή για την Πολιτική Ανάπτυξη και σε άλλες, πολιτικές, και σε άλλες επιτροπές, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερο συντονισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην πολιτική μας. Όσον αφορά το Αφγανιστάν, χρειαζόμαστε αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ Επιτροπής Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Γιατί όσο δεν υπάρχει ένα τέτοιο αποτελεσματικό διάλογο, θα συνεχίσουμε να μην ασκούμε αποτελεσματική πολιτική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τεράστιες δυνατότητες να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος ώστε να αντιμετωπίσουμε τα πολύπλοκα προβλήματα του Αφγανιστάν με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ευχαριστώ. Πολύ, Ευχαριστώ πολύ. Τουλάχιστον να δείξουμε εμεί εδώ το παράδειγμα μια συνεκτική πολιτική. Και τώρα θα ήθελα να ζητήσω εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε τον κύριο Ντέβιτ ή τον κύριο Πόλτα να αναλάβουν το λόγο. Δεν ξέρω αν θέλετε να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε το λόγο. Είναι μια ενδιαφέρουσα έκθεση και προσπαθήσαμε και εμείς να συνεισφέρουμε δίνοντας όσο περισσότερες πληροφορίες μπορούσαμε στον εισηγητή. Πρέπει βέβαια να μπούμε λίγο πιο βαθιά σε αυτά τα θέματα και να μην μείνουμε στην επιφάνεια. Και κυρίω πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη τη δεν είναι σε θέση να καθορίσει το μέλλον και τα όσα θα συμβούν στο Αφγανιστάν. Έχω κάποιε σύντομε παρατηρήσει σχετικά με τη νέα στρατηγική. Βεβαίω υπάρχει μια στρατηγική, την οποία υποστηρίζει η Αφγανική κυβέρνηση και ολόκληρη η διεθνή κοινότητα. Και αυτή είναι η στρατηγική για την ε, Εθνική Ανάπτυξη του Αφγανιστάν 2013 και αυτή θα είναι η βάση για τη θέση του Αφγανιστάν στην διάσκεψη της Καμπούλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε πέρυσι τον Οκτώβριο, όπως αναφέρθηκε, και το οποίο προτίθεται να επιφέρει κάποια λύση σε ένα από τα προβλήματα τα οποία τονίζονται στην έκθεση, δηλαδή στο πρόβλημα της ανεπαρκούς ε, συνεκτικής αντιμετώπισης. Και κάνουμε πρόοδο επ' αυτού, ευτυχώς. Και ως αποτέλεσμα έχει προκύψει και αυτή η γαλάζια βίβλος ε, που είναι διαθέσιμη προς τον εισηγητή και προς οποιονδήποτε ε, άλλο, οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής θέλει να δει πού βρίσκονται, πού πηγαίνουν τα χρήματα της ε, βοήθειας προς τους πολίτες του Αφγανιστάν. Δεύτερον, πρέπει να πούμε ότι είναι δύσκολο να δούμε τον αντίκτυπο. Είναι δύσκολο στο Αφγανιστάν να πούμε ότι έχουμε πάει από το Α στο Β. Καταρχήν γιατί υπάρχουν τεράστια τμήματα της χώρας ε, στα οποία δεν υπάρχει καθόλου πρόσβαση στα χέρια των αντερτών. Είναι δύσκολο να ταξιδέψουμε σε κάποια μέρη της χώρας για πολλούς λόγους. Δεύτερον, εμείς, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, δεν έχουμε επιτόπου επαρκές προσωπικό για να κάνουμε τέτοιου είδους παρακολούθηση. Τρίτον, είναι γεγονός ότι χωρίς ασφάλεια τα εμπλεκόμενα μέρη ε, δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν ε, τα καθιερωμένα δίκτυα πωλήσεως ναρκωτικών. Ε, τέταρτον, χρειαζόμαστε σωστή ασυνόμευση και επιβολή της τάξης σε ολόκληρη τη χώρα για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Και βεβαίως χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των γειτονικών χωρών για την οικοδόμηση του εμπορίου και δεν είναι πάντοτε προφανής η βοήθεια από τις γειτονικέ χώρες πιστεύουμε ε, στο σύστημα διαχείρισης της βοήθειας από την κυβέρνηση όπως έχει καθιερωθεί από την ΕΕ και από την Παγκόσμια Τράπεζα, ε, κάτι το οποίο θα βελτιώσει την παρακολούθηση και προς το παρόν το 50% των όσων κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μέσα από αυτούς τους διάβλους και θέλουμε να αυξηθεί αυτό το ποσοστό. Μπορώ να σα δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία για την πρωτοβάθμια υγεία, για τον αριθμό αγοριών και κοριτσιών στα σχολεία ή για τη βρεφική θνησιμότητα και μπορεί να σα φανούν και καλά αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. Αλλά δεν μπορώ να σα πω με το χέρι στην καρδιά ότι όλα αυτά τα αριθμητικά στοιχεία είναι και σωστά. Παρ' όλα αυτά, έχοντα συζητήσει με πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσει και άλλε οργανώσει που λειτουργούν στο Αφγανιστάν, ε, μπορούμε να πούμε ότι η κάλυψη της πρωτοβάθμιας υγείας είναι σαφώς πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν υπό τους Ταλιμπάν, διότι τότε δεν υπήρχε καθόλου η υγειονομική περίθαλψη. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι καλύπτεται το 80% του πληθυσμού ε, σύμφωνα με την, ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την, τα Ηνωμένα Έθνη και με την Διεθνή Τράπεζα. Και ο, ο των παιδιών στα σχολεία υπολογίζεται γύρω στα 6 εκατομμύρια, ενώ υπό τους Ταλιμπάν ήταν ε, ένα απειροελάχιστο ποσοστό αυτού του αριθμού. Ένα άλλο θέμα τώρα, τα ναρκωτικά, που είναι ένα από τα βασικά προβλήματα. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ε, πιστεύουμε, και αυτή είναι η άποψη της αναπτυξιακής βοήθειας ε, των Ηνωμένων Εθνών, ότι σε κάποιες επαρχίες, σε πέντε επαρχίες είναι περιορισμένο το πρόβλημα των ναρκωτικών και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει βελτίωση στο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες και ιδίως ανάλογα με τις συνθήκες ασφαλείας. Το κέντρο ε, του εμπορίου ναρκωτικών ήταν ε, η, περιοχή Χέλμαν και ακριβώς στην ε, περιοχή Χέλμαν είναι το κέντρο των μαχών αυτή τη στιγμή. Ε, επί τη ευκαιρία να πω ότι η Ρωσία λέει πολλά σχετικά με τα ναρκωτικά, αλλά δεν έχει κάνει και τίποτα για να βοηθήσει, παρά μόνο σε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών εκτό τη χώρα. Ενώ εδώ μιλάμε για το πρόβλημα το οποίο ε, βρίσκεται κατά κύριο λόγο μέσα στη χώρα. Η οικονομική ανάπτυξη είναι ένα σημαντικό θέμα και με ανάπτυξη της γεωργίας και με ανάπτυξη μέτρων ασφαλείας ε, στις περιοχές όπου υπάρχουν πολλοί καλλιεργητές ε, οπιούχων. Και η οικονομική ανάπτυξη είναι ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθούν ε, έσοδα για το Αφγανιστάν, το οποίο συνεχίζει να στηρίζεται απολύτως στη διεθνή βοήθεια. Η αστάθεια και η έλλειψη διακυβέρνησης δημιουργούν διαφορά και όχι το αντίστροφο. Στην έκθεση υπάρχουν ε, ε, διάφορες ε, δυσκολίες οι οποίες εντοπίζονται και για ένα σημείο σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία, ναι βεβαίως είναι σημαντική η επιτευξή ειρήνης για να εκριζωθεί η φτώχεια, αλλά θα πρέπει να επιβάλλουμε και κάποιους όρους επ' αυτού. Δεν αποδεχόμεθα την ειρήνη με οποιοδήποτε τίμημα. Πώς μπορούμε όμως να θέσουμε κάποιες διαχωριστικές γραμμές χωρίς να υπάρχει και επιτόπου κάποια νίκη. Και γι' αυτό ο συνασπισμός προσπάθησε να ακολουθήσει μια δυτή προσέγγιση μέσω του Καρζάη ε, να φτάσει και στους εξεγερθέντες ε, παράλληλα πιέζοντας και ε, τους Ταλιμπάν ε, στην ε, έδρα τους. Μπορούμε να επιτύχουμε πρόοδο χωρίς στρατιωτική δύναμη. Από αυτού δεν έχω ακούσει κάποια απάντηση. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στη γνωστή κατάσταση, δηλαδή ότι κάποια κράτη-μέλη θα αποχωρήσουν μέσα στα επόμενα χρόνια. Ο υπουργός τη Βρετανία έθεσε ένα πενταετές όριο στη στρατιωτική συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο Αφγανιστάν και αυτό το πλαίσιο των πέντε ετών είναι εντελώς διαφορετικό από το πλαίσιο το οποίο γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη ότι είναι απαραίτητο για να επέλθει ανάπτυξη στη χώρα. Σε μια χώρα που βρίσκεται στην κατάσταση του Αφγανιστάν. Η αποτελεσματική διακυβέρνηση είναι η απάντηση και πάλι, αλλά χρειάζονται πολλά χρόνια και πολλή προσπάθεια. Και βέβαια δεν μιλάμε για τον Ιούλιο του 2011. Θα ήθελα να διορθώσω και ένα σημείο παρανόησης ότι έχουμε διακόψει την βοήθειά μας. Δεν έχουμε διακόψει τη βοήθειά μας. Η παρατήρηση αυτή οφείλεται σε μία παρανόηση κάποιου δημοσιογράφου με βάση κάτι που είπε ένας επικεφαλής αντιπροσωπείας στο Αφγανιστάν. Αυτό που είχε πει είναι ότι αποφασίσαμε να περιμένουμε μέχρι ότου καθορίσουμε τη στρατηγική μας για τα επόμενα τρία χρόνια. Το δεύτερο τμήμα του τρέχοντος προγράμματος ανάπτυξης και ε, αυτό ε, να περιμένουμε μέχρι να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα της διάσκεψης Καμπούλ. Δεν μιλήσαμε για διακοπή της παροχής βοήθειας και ε, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, κ. Σάσκας, μαζί με τον κ. Σέντουιλ και με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Αθών, τον κ. Ντεμιστούρα, συνεργάζονται για να επιτευχθεί αυτή η συνοχή που ίσως έλειπε στο παρελθόν μεταξύ των στρατιωτικών. και για την συνοχή της βοήθειας που παρέχεται από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρουμε ότι πολλές από τις παρατηρήσεις ε, και από τα σχόλια που κυκλοφορούν, λέει ο Πρόεδρος, ε, δεν είναι πάντοτε σωστά και είναι καλό που κάνετε αυτή την διόρθωση για να αποκαταστήσετε την αλήθεια. Κύριε Αρλάκη, θα σας δώσω το λόγο για να κλείσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη συζήτηση που έγινε. Για τόσο μεγάλα, τόσο ευρέα θέματα όπως αυτό, ε, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια τόσο εις βάθος συζήτηση. Είναι ε, πολλά τα καυτά θέματα στο Αφγανιστάν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μαζί με το Συμβούλιο είναι τα δύο πολιτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι δουλειά μας να συζητάμε θέματα πολιτικής, μακροπρόθεσμης πολιτικής και να μπαίνουμε στην ουσία των δύσκολων θεμάτων, να μην αποφεύγουμε τις δυσκολίες. Θα προσπαθήσω εν συντομία να απαντήσω στις περισσότερες ερωτήσεις και παρατηρήσεις και θα επικεντρωθώ στα πιο κέρια σημεία. Καταρχήν κύριε Πρόεδρε, η δική σας παρατήρηση για την κρίζωση της παραγωγής παπαρούνας σε χώρες όπου υπάρχει μια εδραιωμένη κυβέρνηση, ενώ στο Αφγανιστάν θα είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι αδύναμη η κυβέρνηση και πολύ ευάλωτη η κοινωνία. Η καλλιέργεια της παπαρούνας έχει καταργηθεί σε όλες τις χώρες, ιδίως σε περιοχές που ήταν εκτός κυβερνητικού ελέγχου. Η καλλιέργεια Παπαρούνα ήταν συγκεντρωμένη ιστορικά σε περιοχέ που ήταν πάρα πολύ δύσκολη η πρόσβασή του. και συνήθω ομάδε ανταρτών ε, διέμεναν σε αυτέ τι περιοχέ και χρηματοδοτούσαν ε, την εξέγερσή του με την καλλιέργεια οπιούχων. Αυτό έγινε πάνω από ένα αιώνα και παρόλα αυτά οι κυβερνήσει με τη βοήθεια τη διεθνού κοινότητα κατάφεραν να πάρουν τον έλεγχο αυτών των περιοχών και να ε, εξαλειφθεί τελικά η καλλιέργεια. Το Πακιστάν είναι το τελευταίο μεγάλο παράδειγμα. Η διεθνή κοινότητα, τα Ηνωμένα Έθνη, χρειάστηκαν 20 χρόνια δουλειά με την κυβέρνηση του Πακιστάν για να εκδηλώσουν την καλλιέργεια οπιούχων στι περιοχέ ε, γύρω-γύρω από το Πακιστάν. Και εγώ ήμουν υπεύθυνο τη παρακολούθηση αυτού του προγράμματο στα τελευταία στάδια του, που δώσαμε τα τελευταία 6 εκατομμύρια δολάρια ε, βοήθεια για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Το Πακιστάν ήταν ε, μεγαλύτερος προμηθευτής, ε, ο οποίου μετά, ε, πριν από το Αφγανιστάν. Πριν από 12 χρόνια θυμάμαι ότι και εγώ είχα προτείνει ένα σχέδιο για την εκδήλωση της παραγωγής οποίου στο Αφγανιστάν. Το σχέδιο αυτό κόστιζε μόνο 25 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Και δεν μπορούσαν να βρεθούν τα χρήματα στη διεθνή κοινότητα για να αρχίσει αυτή η διαδικασία σήμερα με τα τεράστια ποσά που διτίθενται για το Αφγανιστάν δεν είναι πλέον θέμα πόρων. Με τους πόρους που έχουμε μπορούμε να επιχειρήσουμε μεγάλες αλλαγές και ιδίως αυτό για το οποίο συζητάμε στο Αφγανιστάν και μάλιστα σε λιγότερο από πέντε χρόνια, αρκεί να έχουμε το κατάλληλο σχέδιο. Γιατί λέω πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια σημαίνει 20% μείωση της παραγωγής ετησίως, μείωση της αξίας ε, της καλλιέργειας των προϊόντων ε, οποίου που είναι λιγότερο από μισό εκατομμύριο δολάρια το χρόνο. Και μέσα σε πέντε χρόνια θα μπορέσουμε να καλύψουμε την αξία που απαιτείται και το έχω συζητήσει με τους αρμόδιους υπουργούς και κανείς δεν μου είπε ότι είναι μη ρεαλιστικό. Επίσης και οι διεθνείς οργανισμοί πιστεύουν ότι είναι εφικτό. Το ότι υπάρχουν πέντε επαρχίε στο Αφγανιστάν που καλλιεργούν ε, την παπαρούνη είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να επικεντρώσουμε τη δράση μα σε αυτέ τι περιοχέ. Και είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η καλλιέργεια του οποίου στο Αφγανιστάν είναι λιγότερο από 2% της καλλιεργήσιμης επιφάνειας της χώρας. Μην νομίζετε ότι το Αφγανιστάν είναι γεμάτο παπαρούνα που φυτρώνει παντού. Είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της χώρας, το κομμάτι στο οποίο καλλιεργείται η μήκον η πνοφόρος και οι κατάλληλες επενδύσεις από τη διεθνή κοινότητα μπορούν και πρέπει να είναι πολύ αποτελεσματικές. Τώρα, μετά το 2001, σχεδόν για πρώτη φορά ε, το σκεφτόμαστε και είναι σκάνδαλο κατά τη γνώμη μου. 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια δαπάνησαν οι Αμερικανοί για την καταπολέμηση των ναρκωτικών στο Αφγανιστάν με μηδενικό αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν αυτά τα αριθμητικά στοιχεία να τα έχουμε κατά νου για να αποφύγουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει μεγάλη ευθύνη και δεν πρέπει να φοβηθούμε να αναλάβουμε εμεί τον ηγετικό ρόλο, ακόμη και να πούμε στου Αμερικανού, που είναι φίλοι μα, ότι έχουν κάνει τα εξή σφάλματα και να μην ακολουθήσουμε εμεί τα ίδια σφάλματα που έκαναν οι Αμερικανοί στο Αφγανιστάν ή και αλλού. Είμαστε εταίροι, είμαστε φίλοι, αλλά οφείλουμε να πούμε την αλήθεια ο ένα τον άλλον και πρέπει να του βοηθήσουμε, λέγοντά του τι έχουν κάνει λάθο και τι δεν πρέπει να επαναλάβουν στη χώρα αυτή. Η Νικόλ Κινμίσελ τόνισε ε, το θέμα των γυναικών στο Αφγανιστάν. Θα ήθελα να μου δώσει τα στοιχεία σχετικά με τις γυναίκες ε, και αυτά τα οποία έχουμε συμπεριλάβει στην έκθεσή μας για το θέμα των γυναικών ε, ήδη προέρχεται από την Νικόλ και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ δίνοντάς μου τα στοιχεία αυτά για την έκθεση. Πιστεύουμε ότι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των γυναικών πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της ειρηνευτικής διαδικασίας και να μην το θεωρούμε κάτι το ανέφικτο. Επί πολλά χρόνια είχα να κάνω με τους Ταλιμπάν και με άλλους συνομιλητές στο Αφγανιστάν. Όταν έρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και υπάρχουν σαφείς όροι και προϋποθέσεις και γίνεται μια δύσκολη συζήτηση. Αυτά είναι πράγματα που γίνονται. Μην το θεωρήσετε ουτοπία, μην θεωρήσετε ότι είναι κάτι το αδύνατον. Είναι περίεργη χώρα το Αφγανιστάν. Πιστεύω ότι η ενευτική διαδικασία μπορεί να διασφαλίσει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα εφόσον γίνει με το σωστό συντονισμό. Οι Ταλιμπάν γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσουν τον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Είναι γεγονός ε, του οποίου έχουν απόλυτη επίγνωση. Το συζήτησα στην τελευταία μου επίσκεψη στο Αφγανιστάν με κάποιους ε, που πρόσκειται στους Ταλιμπάν και πιστεύουν ότι δεν θα κερδίσουν ποτέ τον ε, πόλεμο και η αποφασιστικότητα της διεθνούς κοινότητας, όπως είπα στην αρχή, είναι τέτοια που δείχνουν ότι μπορεί να μείνουν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως στη Βοσνία, όπως σε πολλές άλλες χώρες και είναι πλήρως ε, μη ρεαλιστικό το να πιστεύουν ότι μπορεί να κερδίσουν. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει και εμείς να πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε εμείς να κερδίσουμε τον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Ήμουν επί τόπου και το συζήτησα με τους στρατιωτικούς, με την ISAF, με όλους τους αρμοδίους και όλοι μου είπαν ότι προετοιμάζουν την ειρήνη στο Αφγανιστάν, προετοιμάζουν τη μεταβατική περίοδο δεν πιστεύουν ότι μπορούν να κυριαρχήσουν στρατιωτικά στη χώρα. Δεν το πιστεύουν εκείνοι. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος να το πιστεύουμε εμείς. Για το θέμα ε, που έθεσε ο κύριος ε, Πρέντα, για τις παρατηρήσεις του κύριου Πρέντα. Αυτός ο τίτλος «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης» δεν ξέρω ε, γιατί ε, δεν υπάρχει πια. Ε, αρχικά έλεγε στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το επαναφέρουμε, να λέει στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Αφγανιστάν. Γιατί επ' αυτού ακριβώς πρόκειται. Αυτό προσπάθησα να κάνω, να δω ποια είναι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν και να αναπτύξω κάποιες ιδέες για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Άρα είναι κάτι το οποίο πολύ εύκολα μπορεί να διορθωθεί αυτό που παραθέσατε από τον Καρλ Μπίλντ, άκουσα εγώ ε, την ηχογράφηση της ομιλίας ε, του Καρλ Μπίλντ ε, και σημείωσα ακριβώς αυτά τα οποία είχε πει στην τελευταία συνάντηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων εδώ. Όσον αφορά τους Ταλιμπάν, δεν νομίζω ότι είμαι ιδιαίτερα γενναιόδος. Αυτό που λέω σε αυτό το κεφάλαιο, αυτό που λέω για την εκρίζωση της καλλιέργειας ε, Παπαρούνας, είναι το εξή. Λέω ότι τα Ηνωμένα Έθνη υποχρέωσαν τους Ταλιμπάν ε, να απαγορεύσουν την καλλιέργεια. Και το ήμουν εγώ ο ίδιος υπεύθυνο και σας διαβεβαιώνω ότι χρειάστηκαν πέντε χρόνια για να απομονώσουμε καταρχήν πολιτικά τους Ταλιμπάν τους Ταλιμπάν και τους φίλους τους Πακιστάνους και Τουρκμένισταν, να τους απομονώσουμε από πολιτικής πλευράς και όταν είδαν ότι ήταν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους, άρχισαν ε, να προσέχουν περισσότερο. Είχαν ε, κυρώσει των Ηνωμένων Εθνών εναντίον τους και τη δεύτερη φορά των κυρώσεων αποφάσισαν ε, να αποδεχθούν την απαγόρευση της καλλιέργειας, την οποία τους, είχε επιβάλει, τους είχαν επιβάλει τα Ηνωμένα Έθνη. Και όταν μπήκαν οι Αμερικανοί στην Καμπούλια χρόνια αργότερα, δεν υπήρχε καλλιέργεια οποίου χάρη στην δράση των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν κάτι το οποίο είχε επιτυχία στο τέλος. Και μια παρόμοια δράση σήμερα με τους τεράστιους πόρους που διαθέτουμε και με πολύ μεγαλύτερη πολιτική πίεση δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην έχουμε το ίδιο θετικό αποτέλεσμα. Με συνομιλητές που είναι πολύ πιο συζητήσιμοι από ότι οι Ταλιμπάν εκείνη την εποχή δεν σας αρέσει η παράγραφος 59 ε, σχετικά με τον Μπούς και λοιπά, ε, είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε. Δεν έχω πρόβλημα να το αλλάξω αυτό, να αλλάξω αυτή την παράγραφο που δεν είναι ουσιαστική. Τα ειθνικά στοιχεία για το κόστος του πολέμου για την εξάλληψη της φτώχειας στο Αφγανιστάν που κοστίζει πέντε μέρες πολέμου ίσως είναι υποτιμημένα γιατί τώρα έχουμε τα τελευταία στοιχεία που έχει δώσει το Κογκρέσο για το κόστος του πολέμου στο Αφγανιστάν και αν τα ξαναέγραφα τώρα αυτά που γράφω θα έλεγα ότι λιγότερο από πέντε μέρες πολέμου θα αρκούσαν για να εξελιχθεί η καλλιέργεια της Παπαρούνας. Και χθε ε, έγινε μια συζήτηση στο Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου το Πεντάγωνο είπε ότι ένα γαλόνι βενζίνης στο Αφγανιστάν κοστίζει 400 δολάρια. Το να παραδοθεί αυτή η ποσότητα πετρελαίου στο στρατό που βρίσκεται στο Αφγανιστάν. Αυτό μας δίνει μια εικόνα των απαιτήσεων για τη διατήρηση των στρατευμάτων στο Αφγανιστάν. Πρέπει να τα λάβουμε υπόψη αυτά τα στοιχεία για να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή εικόνα της κατάστασης στο Αφγανιστάν και της απόσυρσης από το Αφγανιστάν. Εγώ επικεντρώνω το ενδιαφέρον μου στην ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εσείς θέλετε να προσθέσουμε και κάποιες άλλες παρατηρήσεις, είμαι ανοιχτό. Μπορούμε να προσθέσουμε και κάτι παραπάνω για να κινηθούμε προς την κατεύθυνση που εσείς επιθυμείτε. Για τις παρατηρήσεις του κυρίου Νόιζε από την ομάδα των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για τη διάκριση στρατιωτικής και μη στρατιωτικής βοήθειας, συμφωνώ. Πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση. Παρότι πρέπει να πω, ενώ συμφωνώ απολύτως μαζί σας, ε, οφείλω να πω ότι είδα ε, το πώς δίδεται η Ιταλική βοήθεια στο Αφγανιστάν, στο Χεράτ. Και εγώ δεν είμαι υπέρ του να, παραδει... να δίνετε στρατιωτική βοήθεια, αλλά πρέπει να σας πω ότι το καλύτερο παράδειγμα που έχω δει στο Αφγανιστάν ήταν αυτό. Ήταν η μοναδική περίπτωση που υπήρχε ένα πρόγραμμα σωστό, χωρίς πατάλη, χωρίς ε, διαφθορά, με αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις οργανικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν κλπ. Δεν λέω ότι είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε. Θα ήθελα τα χρήματα να διακινούνται από μη στρατιωτικές, ε, από μη στρατιωτικούς διάβλους, αλλά υπάρχουν και ε, λόγοι για τους οποίους θα μπορούσαμε ε, να υποστηρίξουμε και αυτή τη βοήθεια από τους στρατιωτικούς. Επίσης, Συμφωνώ με την ιδέα σας ε, του να συμπεριλαμβάνονται και οι περιφέρειες, ε, η, όλη περιφέρεια, το Πακιστάν, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα. Πιστεύω ότι είναι μια άλλη εναλλακτική λύση για την επίλυση της κρίσης στο Αφγανιστάν. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, έχουν μεγάλα συμφέροντα στο Αφγανιστάν και πολλές ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε αλλά αν χάσουμε την βοήθεια από την ε, συνολική περιφέρεια, ε, αν αφήσουμε απ' έξω τη βοήθεια από την περιφέρεια, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τη σωστή τελική λύση για το Αφγανιστάν. Πρέπει να ε, συμμετάσχουν και οι χώρε τη περιφέρεια. Δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε την κατάσταση στο Αφγανιστάν στο τέλο τη δεκαετία του 90, όπου το Αφγανιστάν ήταν πεδίο μάχη με στρατούς και ομάδες που χρηματοδοτούνταν από όλες τις χώρες της περιφέρειας. Κάποιους χρηματοδοτούσαν χρηματοδοτούσε το Ιράν, κάποιους η Ρωσία, κάποιους ε, οι Αμερικανοί, κάποιους ε, οι Ινδοί που έπαιζαν το παιχνίδι τους, ε, Πακιστάν, Ταλιμπάν κλπ. Δεν το έβαλα αυτό το θέμα στην έκθεση, ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. και μπορεί να μας οδηγήσει σε διαφωνίες. Πρέπει να αποφύγουμε την παρεμβολή στις εσωτερικές υποθέσεις του Αφγανιστάν από τις χώρες της περιφέρειας και δεν θα πρέπει ε, να διαχειριζόμαστε εμείς την πολιτική του Αφγανιστάν και θέλουμε να αποφύγουμε ε, την κατάσταση του τέλους της δεκαετίας του 90 με την παρέμβαση όλων των γειτονικών χωρών. Κύριε Μέγερ, συμφωνώ και με αυτή τη δική σας πρόταση για το ότι πρέπει να συμμετέχει η γενικότερη περιφέρεια και η πρόσφατη δήλωση ε, του νέου επικεφαλής ε, από πλευράς των ΗΠΑ δεν είναι πάρα πολύ χρήσιμη, διότι υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι είναι δυνατή μια στρατιωτική λύση στο Αφγανιστάν και τώρα αρχίζει αυτή η μη δηλωμένη ε, στρατιωτική προσέγγιση ε, για την ε, εξάλληψη των επικεφαλής των ανταρτών και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη διεθνούς στρατηγικής που εξέτασε ιστορικά 300 ε, περιστατικά ε, όπου δυνάμεις κατοχής προσπάθησαν να αποκεφαλίσουν την ηγεσία των ανταρτών και μόνο στο 7% των περιπτώσεων επέτυχαν τέτοιες ε, στρατηγικές, το 93% απέτυχαν. Συμφωνώ και με τον κύριο Γκέρενς ότι πρέπει να γίνει μια διάκριση ε, για το είδος της διαφθοράς που υπάρχει στο Αφγανιστάν και οποιαδήποτε μελλοντική βοήθεια στο Αφγανιστάν, ακόμη και αν αυξήσουμε τη βοήθεια που διακινείται μέσω της κυβέρνησης, θα πρέπει η βοήθειά μας να συνοδεύεται από κατάλληλα μέτρα ελέγχου. Έχω σημειώσει τις παρατηρήσεις του κυρίου Μάουρο για τη διεθνή βοήθεια και συμφωνώ μαζί σας σε μεγάλο βαθμό, ότι πρέπει να βρούμε το κατάλληλο μείγμα διάβλων παροχής βοήθειας. Πάντως, οπωσδήποτε, πρέπει να αυξήσουμε το ποσό που διακινείται μέσω της κυβέρνησης του Αφγανιστάν. Ήδη διακινείται το 50% της βοήθειας μέσω της κυβέρνησης, ζήτησε 80% η αφγανική κυβέρνηση χθε και συμφωνώ ότι περισσότερα χρήματα θα πρέπει να περνούν από το διάβλο της κυβέρνησης. Διότι αν θέλουμε να έχουμε μια ε, κυβέρνηση νομιμότητας θα πρέπει να τονίσουμε ναι, ακριβώς το ότι η δική μας βοήθεια περνάει από την κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Δεν είμαι υπέρ καμιάς αύξηση ε, ιδιωτικών ε, παραστατιωτικών ομάδων, ούτε ιδιωτικών μονάδων και συμβαλωμένων θα πρέπει μέσω της κυβέρνησης να περνάει για να διακοπεί η κατάσταση που τροφοδότησε τον εμφύλιο πόλεμο επί δεκαετίες. Δεν μπορώ να μπω σε πολλές λεπτομέρειες για τα τελευταία θέματα που έχω σημειώσει. Συμφωνώ με τη συνεργασία με το Κογκρέσο και έχουν έρθει επαφή μαζί μου κάποιοι Αμερικανοί βουλευτές που ενδιαφέρονται ακριβώς για το ίδιο θέμα και πριν από λίγες μέρες μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, αυτή που σα δείχνει η Warlord Inc., κατατίστηκε από το Κογκρέσο, από την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Εξωτερικών Υποθέσεων και είναι μια έκθεση που μας βοηθάει να κατανοήσουμε το πρόβλημα της διεθνούς βοήθειας στο Αφγανιστάν και τι ακριβώς πρέπει να αλλάξει. Μια τελευταία παρατήρηση προς τον κύριο Τιερ. Δεν συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη της δεν μπορεί να προσδιορίσει το μέλλον του Αφγανιστάν. Και βέβαια δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει τα πάντα στο Αφγανιστάν. Αλλά το Αφγανιστάν αποτελεί μια μεγάλη αποτυχία της διεθνούς πολιτικής και της πολιτικής των ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει λόγο και μπορεί να αναλάβει και τον ηγετικό ρόλο με νέες ιδέες, με νέα στρατηγική σε φιλικό περιβάλλον, γιατί οι Αμερικανοί είναι φίλοι μας όπως ήδη είπαμε. Αλλά έχουμε εμείς μεγάλη ευθύνη στο Αφγανιστάν. Έχουμε στρατεύματα, η κοινή γνώμη ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το θέμα. Δεν πρέπει να ακολουθήσουμε απλώς τους Αμερικανούς και να επαναλάβουμε τα σφάλματά τους. Και αυτόματος ε, ζητούν και πολλοί Αμερικανοί. Μα ζητούν οι Αμερικανοί να τους βοηθήσουμε να αλλάξουν την πολιτική τους στη χώρα. Και ο Ομπάμα προσπαθεί να αλλάξει την προηγούμενη πολιτική Μπούς, επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλη ευθύνη επί του θέματος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να επισημάνω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 7η Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα. Θα ζητήσω από τον κύριο Παντζέρη, αν θέλει να μας παρουσιάσει το θέμα. Έκθεση σχετικά με την κοινή αντιπροσωπεία αφεντεύε Budget. Επίσκεψη στη Μέση Ανατολή το Μάιο του 2010. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σημείο στην ημερήσια διάταξη προβλέπει λιγάκι τον απολογισμό της επίσκεψης που έγινε στην Ιερουσαλήμ και στη Γάζα. με τα μέλη των τριών επιτροπών. Της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης και Προπολογισμών. Η επίσκεψη αυτή, πέρα των ε, διεξεφισμών που την συνόδευσαν, ήταν πολύ σημαντική. Διότι μπορέσαμε να συναντηθούμε και με τις αρχές του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Ήταν μια επίσκεψη που επέτρεψε να κατανοήσουμε επιτόπου πώς έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Όπως γνωρίζουμε λίγο πολύ όχι. Στόχοι της επίσκεψης ήταν οι εξής τρεις. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η ανθρωπιστική βοήθεια, η χρήση των κονδυλίων που εκταμιεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την περιοχή και να δούμε πώς πάει η πολιτική διαδικασία, η ειρηνευτική διαδικασία. Είχαμε σημαντικές συναντήσεις και στην Ιερουσαλήμ και στη Ράμαλα και στην Χευρώνα και στην ε, Ναμπλούς και επισκεφθήκαμε και τη Γάζα. Και αυτό χάρη στην Αίγυπτο και όχι στο Ισραήλ. Οι συναντήσεις που είχαμε ήταν ιδιαίτερα σημαντικές και καταφέραμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Καταγράψαμε το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρά το μεγάλο πρόβλημα της χρήσης του στην Γάζα. Όμως υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθούμε συνεχώς αυτή την κατάσταση και ως προς την ανθρωπιστική βοήθεια. Είδαμε ότι για τη δυτική όχθη συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα, περισσότερο όμως στη λωρίδα της Γάζας και για την ειρηνευτική διαδικασία Είδαμε στην πράξη ποιες είναι οι δυσκολίες και των έμεσων διπλωματεύσεων και των προβλημάτων στις σχέσεις μεταξύ της Παλαιστινικής Αρχής και των Ισραηλινών Αρχών. Όλοι βεβαίως εκφράσαμε την ευχή η κατάσταση αυτή να απεμπλακεί. Και μετά τη συνάντηση που έγινε στο Λευκό Οίκο μεταξύ Ομπάμα και Νετανιάχου. Τώρα και στην Κνέσετ, στη συνάντησή μας με τις Ισραηλινές Αρχές και με τους ίδιους τους πολιτικούς ευθύνοντες, ανέκυψε ένα σημαντικότατο ζήτημα που συνεχίζει να βρίσκεται με τρόπο σχεδόν ε, επίμονο το θέμα της ασφάλειας, το θέμα της ασφάλειας του Ισραήλ. Αυτό ανακύπτει συνεχώς τις συζητήσεις μας. Πιστεύω ότι είναι ένα ζήτημα που και εμείς θα πρέπει να το αναλάβουμε ως ευθύνη και να το εξετάσουμε διότι εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει επαρκής γνώση ότι το θέμα της ασφάλειας σχετίζεται άμεσα με το κατά πόσο θα προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία αν δεν, κατα... αν δεν οι εντάσεις για τα ζητήματα ιδίως που εντοπίζουμε όπως η πολιτική επικισμού ιδίως στην Δυτική στην Ανατολική Μάλλον Ιερουσαλήμ, το θέμα της Λωρίδας της Γάζας και ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων, κάτι που εξέταζε εκείνο το διάστημα που πήγαμε εμείς, η Κνέσετ. Επίσης, έπρεπε να εξηγήσουμε τους λόγους που είχαμε να παροτρύνουμε την πρόοδο της νευτικής διαδικασίας προβάλαμε το επιχείρημα ότι αυτό θα προάγει και την ασφάλεια του Ισραήλ. Όμω, για να έχουμε καλύτερη γνώση του θέματο, και νομίζω ότι αυτό το πετύχαμε με την επίσκεψή μα, πρέπει να δούμε τι δηλώσει κάνουμε και στι συναντήσει που έχουμε. Και τα επιχειρήματά μα θα είναι πιο ισχυρά αν έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η πολιτική δράση και ενεργό συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην ειρηνευτική διαδικασία δεν γίνεται ιδιαίτερα κατανοητή και ιδιαίτερα υπό το φως, της συμμετοχής της ε, οικονομικής που έχουμε, της ανθρωπιστικής ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να φοβάται να θέσει και τους δικούς της όρους είτε στις χώρες της περιοχής αλλά και στον, ε, στο σύνολο του κουαρτέτου και ιδίως στην άρση του αποκλεισμού στους, ε, στους καταβλισμούς στην Δυτική Ιερουσαλήμ, στο ρόλο που διαδραματίζουν οι χώρες της περιοχής, πρέπει όλοι να συνεισφέρουν στην ειρηνευτική διαδικασία και στην αναθεώρηση της δικής μας της συμμετοχής ως Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να περάσουμε σε άμεσες πλέον, απευθείας διαπραγματεύσεις, να αφήσουμε το στάδιο των ατύπων διαπραγματεύσεων. Από την επίσκεψη λοιπόν αυτή διεφάνει η ανάγκη να αναλάβει έναν ενεργότερο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς στις δηλώσεις που τόσο συχνά κάνουμε. Μία προσωπική μου άποψη να εκφράσω εδώ. Δεν μπορούμε να επιμένουμε στο ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την αρχή της δημοκρατίας, όπως κάναμε στην Παλαιστίνη και με τις εκλογές, με τις, μάλλον με τις ευχές που διατυπώθηκαν και τις εκλογές που οργανώθηκαν, εκεί είδαμε να κερδίζει η Χαμάς. Όμως υπήρξε κράτηση πολλών βουλευτών και σιωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά απέχουν πολύ από τις στυλώσεις μας. Δηλαδή, από τη μια λέμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε έναν δρόμο και μετά δεν αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει ισχυρή παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν διευκολύνει καμία δημοκρατική διαδικασία. Ούτε δημιουργεί προποθέσει ευνοϊκέ για τη δημοκρατία. Δημιουργεί δυσχερεί συνθήκε. Η επίσκεψη λοιπόν, όπω είπα, ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Τέθηκε στην ημερήσια διάταξη και το θέμα τη ε, ε, ελαφριά αλλαγή πορεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση διότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να έχουμε συνεχώς κατά νου την επίσκεψη αυτή και να ενισχύσουμε και τη σχέση μεταξύ των τριών ε, επιτροπών, των κοινοβουλευτικών επιτροπών που συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία. Επίσης, σημαντικό θα ήταν να αναλάβει ενεργότερο ρόλο η ομάδα που δημιουργήσαμε στο Κοινοβούλιο για τα θέματα της Μέση Ανατολή με την προεδρία του κ. Πέτερινγκ γιατί νομίζω ότι έτσι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε πιο συγκεκριμένα κάποιου στόχους από την πλευρά τουλάχιστον του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Πέτσερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμμετείχα ως πρόεδρος στην αντιπροσωπή αυτή, όπως είπε και ο κύριος Παντσέρη, πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τη Μέση Ανατολή. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τον κύριο Παντσέρη που ηγήθηκε της ε, αποστολής. Έχω την εντύπωση ότι σε τέτοιου είδους αποστολές και είναι πολλοί παρόντες από που ήρθαν μαζί μας, πρέπει να έχουμε ένα στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Λύση δύο κρατών Ισραήλ με ασφαλή σύνορα και Παλαιστίνη με ασφαλή σύνορα. Και εδώ αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ ήθικο, πλαστικό ή πολύ μεγαλόστομο και φιλόδοξο, αλλά είναι η ουσία και ο πυρήνας του προβλήματος. Η αξιοπρέπεια ενός Ισραηλινού είναι ακριβώς η ίδια με την αξιοπρέπεια ενός Παλαιστινίου. Και τούμπαλιν, ο Παλαιστίνιος έχει ακριβώς την ίδια αξιοπρέπεια με τον Ισραηλινό και θα πρέπει να έχει την ίδια μεταχείριση. Αν θέλουμε λοιπόν τη λύση αυτή των δύο κρατών, έχουμε την εντύπωση ότι κάποιοι εκατέρωθεν όμως δεν επιθυμούν δύο κράτη. Κάποιοι στο Ισραήλ και είδαμε χτες καταστράφηκε πάλι ένα σπίτι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ένα Παλαιστινιακό. Βλέπουμε επικισμούς από το Ισραήλ και διώχνουν από τις αιστείες τους Παλαιστινίους. Ε, αυτό είναι ε, αντιφατικό με τα δύο κράτη. Το ίδιο κάνει και η Χαμάς όταν στέλνει ρουκέτες από τη λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ. Δηλαδή και στις δύο πλευρές υπάρχουν άνθρωποι που δεν επιθυμούν ούτε την ειρήνη ούτε τη λύση των δύο κρατών και θέλουν να την αποτρέψουν. Και κάτι που με ενόχλησε. Κάποιοι κατηγορούν την ίδια τους την κυβέρνηση ότι είναι το ε, ε, μάλλον όταν κάποιο επικρίνει την Ισραηλινή κυβέρνηση σε κατηγορούν ότι είσαι στο αντιισραηλινό λόμπι. Όταν επικρίνει τη Χαμάς δεν είσαι αντιπαλαιστινιακό λόμπι. Δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Και σε ό,τι αφορά τη Γάζα και τα θλιβερά γεγονότα πριν από λίγε εβδομάδες έδειξε ότι η κοινή γνώμη απέκτησε και πάλι συνείδηση του προβλήματος. Και φαίνεται ότι θα ανοίξει λίγο η Γάζα. Ένα τμήμα της δικής μας αντιπροσωπείας, όπως είπε ο κ. Πανσέρη, αναγκάστηκε να πάει μέσω Αιγύπτου. Νομίζω ότι ο συνάδελφος Κράισερ Ντόφρερ ήσασταν εκεί. Όχι, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι αναγκάστηκαν να πάνε από την Αίγυπτο. Τελαβίβ Κάιρο, η Βερονίκ Ντεκεζέρα, ας πούμε. Ε, είδα ότι ήταν πέταξαν, μάλλον ε, πήγαν Τελαβίβ Κάιρο και μετά από το Κάιρο με το λεωφορείο στη Ράφα, στο πέρασμα, για να πάνε στη Γάζα. Και ακούσαμε και τον κύριο Φαγιάτ. Τι σημαίνει διατήρηση ε, του αποκλεισμού. Δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά σχολείο. Δεν μπορούν να χτιστούν τα κτίρια που έχουν καταστραφεί. Και οδηγείται σε απομόνωση ε, η Γάζα και τελικά αυτό είναι νερό στο μήλο της Χαμάς. Όποιο θέλει να διατηρηθεί το εμπάργο και αποκλεισμό στη Γάζα βοηθάει τη Χαμά. Δεν μπορούμε να έχουμε εμεί τέτοιο στόχο. Λοιπόν, καθήκον μα είναι ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με την Αμερική, μαζί με την τετραμερή, όπω είπε και ο συνάδελφο Παντσέρη, το λεγόμενο κουαρτέτο, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουν οι επικισμοί και η αντίστοιχη πολιτική. Και αν σταματήσει και ο αποκλεισμό τη Γάζα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται όμω ότι δεν θα περνάνε όπλα στη Γάζα για να γίνονται επιθέσεις και βομβαρδισμοί ε, στο Ισραηλινό έδαφος. Και η κριτική μας ε, απευθύνεται σε εκείνους που οξύνουν τα πνεύματα και σε κάποιους θερμοκέφαλους και στις δύο πλευρές. Τελευταία παρατήρηση. Αν διατηρεί τη δέσμευσή του ο πρόεδρο Ομπάμα για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, τότε θα πρέπει να κάνουμε εμεί ό,τι μπορούμε για να το υποστηρίξουμε. Και είμαι βαθύτατα πεπισμένο, χωρί δυνάμει ασφαλεία τη διεθνού κοινότητα, δεν ξέρω ποιοι θα είναι, ο ΙΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, α το δούμε αυτό. Α τα αφήσουμε ανοιχτό. Αλλά αν δεν υπάρξουν ε, δυνάμει ασφαλεία ε, στη Μέση Ανατολή όπου να συμμετέχουμε κι εμεί, δεν ε, είναι δυνατή η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, κατά την άποψή μου. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε και να είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε. Και κατά την άποψή μου, και τελειώνω με αυτό, στη Μέση Ανατολή διακυβεύονται πολύ περισσότερα από την ειρήνη Ισραήλ-Παλαιστίνης, όσο σημαντικό και είναι αυτό. Αν δεν υπάρξει εκεί η ειρήνη, αυτό θα έχει επιπτώσει στη σχέση μα με το σύνολο του Ισλαμικού και του Αραβικού κόσμου και την Ένωση για τη Μεσόγειο. Μπορούμε να την ξεχάσουμε την Ένωση για τη Μεσόγειο, δεν κάνουμε πρόοδο ε, στις σχέσεις Ισραήλ-Παλαιστίνης. Γι' αυτό είπαμε διακυβεύονται πολύ περισσότερα, πάρα πολύ περισσότερα από τα δύο κράτη και μόνο και μας συνιστώ σε όλου μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας εδώ αλλά και στην Ομάδα Εργασίας για τη Μέση Ανατολή να διατηρήσουμε τη συγκέντρωσή μας στη Μέση Ανατολή και να υψώσουμε τη φωνή μας. Και αν θεωρούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι κάνει κάτι στραβό η Παλαιστίνη, η Χαμάς, η Ισραηλινή κυβέρνηση, θα το λέμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να το λέμε και δεν θα πρέπει να ακούμε τέτοιες αιτιάσεις και ύβρις ότι είμαστε μονομερείς. Όχι, δεν είμαστε ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Θέλουμε να υποστηρίξουμε την ειρήνη αυτό που είδαμε και στην Ευρώπη μετά το 1945 με το σχέδιο του Σούμαν και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αν υπάρχει καλή βούληση θα μπορούσε αυτό να γίνει πραγματικότητα και στη Μέση Ανατολή. Και να μην μας λένε ότι είναι όλα αυτά οράματα. Γιατί στην Ευρώπη αυτό να έγινε πραγματικότητα και να μην μπορεί να γίνει αλλού. Βέβαια όταν υπάρχει καλή βούληση επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ κύριε Πέτρινγκ ή Βερονίκ Ντεκεζέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον συνάδελφο Πανσέρη και τον Πρόεδρο κύριο Πέτερη. Όταν λέει ο κύριος Πέτερινγκ ότι η αξιοπρέπεια ενός Παλαιστινίου θα πρέπει να ταυτίζεται με την αξιοπρέπεια ενός Ισραηλινού, πρέπει να προσθέσουμε και η ασφάλεια ενός Ισραηλινού θα πρέπει να είναι ίδια με την ασφάλεια ενό Παλαιστινίου. Και πάει λέγοντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πολύ δύσκολο να το λέμε. Δεν μιλάμε για ίσες αποστάσεις, μιλάμε για ίσα δικαιώματα. Έχουν το δικαίωμα όλοι οι άνθρωποι να ζήσουν μια ζωή με ελπίδες, με εκπαίδευση, με δυνατότητα να κυκλοφορούν. Από τη μια στο όνομα της ασφάλειας του Ισραήλ που δεν είναι και καλό αυτός ο υπολογισμό μακροπρόθεσμα. Λοιπόν, στο βωμό τη ασφάλειας του Ισραήλ τι να κάνουμε, λυπούμεθα κτλ. αλλά όλα τα άλλα πάνε περίπατο. Όχι, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη λογική ως Ευρωπαίοι. Και συμφωνώ με τον κύριο Πέτερινγκ να έχουμε ένα όραμα για δικαιώματα και να βρούμε λύσεις που να εξασφαλίζουν και να εγγυώνται τα δικαιώματα όλων και μόλις ε, τα πούμε αυτά τα πράγματα μας κατηγορούν και μας συμβρίζουν. και είναι πάρα πολύ οδυνηρά όλα αυτά. Ήθελα να πω κάτι άλλο. Είχα πάει με μια αντιπροσωπεία υπό την ηγεσία της Εύα Ζολή στη Γάζα και άλλοι, κυρία ε, και κάποια άλλα μέλη. Πάρα πολύ σύντομα για όσους δεν είχατε την ευκαιρία να ενημερωθείτε, η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας ποια είναι. Γιατί θα έρθουμε στη συνέχεια στη χρηματοδότηση, στο πρόβλημα αυτό. Έχω πάει πολλές φορές στη Γάζα από την ε, ε, περασμένη επιχείρηση είχα να πάω και η κατάσταση είναι ε, τρομακτική. Η μαύρη αγορά στα τούνελ έχει λάβει τώρα διαστάσεις πραγματικά επιχειρηματικές ολοκένουργια φορτηγά που έχουν φτάσει σε ανταλλακτικά μέσα από τα τούνελ, είναι στην έξοδο των τούνελ και παίρνουν τα ε, εμπορεύματα και τα πουλάνε, τα πηγαίνουν στα μαγαζιά. Και τσιμέντο έχουν ε, αλλά το 90% των κατοίκων της Γάζας δεν μπορούν να κερδίσουν τίποτα από αυτή τη μαύρη αγορά. Ζουν από κάποια επιδόματα, από μια δημόσια ελεημοσύνη και ε, αγωθά υπάρχουν, τα βλέπουν στα μαγαζιά αλλά δεν μπορούν να τα αγοράσουν και αυτό δημιουργεί τεράστιες εντάσεις, απογοητεύσεις και προβλήματα. Και είναι ε, έτσι η κατάσταση. Ε, αυτός ο αποκλεισμός είναι τελείως αντιπαραγωγικός γιατί ε, στοχεύει τον πληθυσμό που δεν πρόσκειται στη Χαμάς. Η Χαμάς έχει και τσιμέντο και λεφτά και χτίζει τζαμιά, σχολεία με και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά εκείνοι που δεν έχουν τα στοιχειώδη και δεν βρίσκονται και κοντά στη Χαμάς είναι τελείως άπο. Και το κράτος και η Ούνρα ε, του ΟΗΕ δεν μπορεί να αγοράσει εντός αγωγικών μαύρο τσιμέντο από τη μαύρη αγορά και όλα τα υλικά που υπάρχουν αλλά είναι προϊόν μαύρη αγοράς και βρίσκεται και εκείνη σε δενή θέση και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και μας λέει η Ούνρα λοιπόν ότι δεν μπορεί να δώσει παρά μόνο τη μισή μερίδα ε, θερμίδων που είναι απαραίτητη για την επιβίωση. Και όταν μα λένε ότι δεν υπάρχει ανθρωπιστικό δράμα στη Γάζα, εγώ απαντώ, εκείνοι που τα λέγουν αυτά δεν έχουν πάει στη Γάζα σίγουρα. Και... Εντάξει, παραδέχομαι, δέχομαι να πιστέψω ότι δεν είναι και ενήμεροι. Αν δεν σταματήσει απολύτως ο αποκλεισμός, αν δεν αρθεί τελείως με δυνατότητες εξαγωγών, δηλαδή μια ανάπτυξη της οικονομίας, προς το εξωτερικό μια διεθνούς οικονομία ή ακόμα και μια οικονομία από τη Γάζα προς τη δυτική όχθη. Εάν δεν υπάρχουν αυτά ε, και όσο δεν υπάρχουν είναι απολύτως απαραίτητη βοήθεια. Εκτός από εκείνους προνομιούχους όπως είπαμε που είναι περί τη και δεν τα έχουν ανάγκη αυτά. Και όταν άκουσα στην ομάδα εργασίας ε, τους εκπροσώπους και χτες το βράδυ το Σαλάμ Φαγιάτ μας λένε ότι λυπούμεθα πάρα πολύ, αλλά μας χρειάζονται ακόμα αυτά τα χρήματα. Γιατί ε, εφόσον δεν είναι πλήρη η σιάση του αποκλεισμού, είναι σταγόνα στον ωκεανό αυτό που προτείνει το Ισραήλ. Εντάξει, ας το καλωσορίσουμε τι προτείνει, γιατί κάθε βήμα προς τα εμπρός είναι αξιόλογο και αξιέπαινο, αλλά δεν θα αλλάξει την κατάσταση. Τι προτείνει λοιπόν να μπει Κάποια αγαθά για την ανοικοδόμηση των υποδομών, ας πούμε, και των έργων της Ούντρα, αλλά αυτό καλύπτει μόλις το 5% των αναγκών από πλευρά σχολείων, υποδομών, κτηρίων κτλ. Ενώ ο πληθυσμός περιμένει, τα παιδιά μεγαλώνουν, 80% του πληθυσμού της Γάζας είναι ιδιαίτερα νέοι και δεν έχουν άλλες εναρκτικές λύσεις παρά να πάνε στα ε, θρησκευτικά σχολεία της Χαμάς. Δυστυχώ θα πρέπει να εξακολουθήσουμε την πίεση και να εξακολουθήσουμε να τους υποστηρίζουμε στις ανάγκες τους οικονομικά. Ε, λυπούμαστε γι' αυτό. Και εκείνοι να δείτε πόσο λυπούνται. Είδαμε επιχειρηματίες στη Γάζα, οι οποίοι θέλουν να εργαστούν, θέλουν ε, να ασχοληθούν με το εμπόριο, νερό έχουν υπόγειο και θερμοκήπια για να μπορούν να καλλιεργήσουν. Θέλουν να δουλέψουν οι άνθρωποι, αλλά ε, είναι δεμένα τα χέρια τους. Αλλά τα θερμοκήπια είναι άδεια, δεν παράγεται τίποτα. Γιατί και να παράγουν να τα αφήσουν να σαπίζουν μέσα στη γάζα αφού δεν μπορούν να βγουν τα εμπορεύματα. Τι να τα κάνουν. Γι' αυτό, γιατί κάθεστε τόσο πίσω εκεί. Πόσο προβλέπετε 20 εκατομμύρια ευρώ για την Ούνρα. Αρκούν αυτά γιατί ο Τζέγκινγκ ε, τα υπολογίζει ε, σε 100 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ ανισχυτικά αυτά. Και το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φέρουμε αντιμέτωπη την ούρα με το Σαλάμ Φαγιάτ αρκούν αυτά τα χρήματα, γιατί είστε τίμιος και ειλικρινής και είμαι βέβαια ότι θα μου απαντήσετε. Not, not now. Ναι, αλλά όχι τώρα, λέει ο Πρόεδρος, διότι μπορεί να υπάρξουν και άλλες ερωτήσεις. Τελειώσατε, κύριε Δεκεζέ. Χωρίς μικρόφωνο. Ναι, κάνω την ερώτηση και περιμένω απάντηση. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι Έχουμε και το διευρυμένο προεδρείο που πρέπει να συνδυάσει μετά, έτσι. Και θα σας παρακαλούσα να κλείσει εδώ ο κατάλογος των ομιλητών. Έχουμε ήδη. Πώς. Έξι. Και η ώρα είναι αυτή που είναι, 11.30. Η κυρία Κυρνίλσεν και μετά ε, θα σας παρακολουθώ να επικεντρωθείτε σε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παντζέρη που έκανε μια πολύ καλή έκθεση και ακούσαμε αυτά τα οποία είδαμε και νιώσαμε κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης και αυτά που είπε η κυρία Βερονίκτα Κεζέρ, ε, ήμουν και εγώ μαζί της στην ε, Γάζα. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω λοιπόν όλα αυτά. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια σημεία. Όταν μιλάμε για αξιοπρέπεια, ο κ. Πέτερινγκ πολύ σωστά ανέφερε την αξιοπρέπεια των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών. Θα ήθελα να υπενθυμίσω την ευθύνη μας ε, ημών ως Ευρωπαίων για το θέμα της εισαγωγής προϊόντων που ξεκινούν από, τις, από τα κατεχόμενα, γιατί η ε, αξιοπρέπεια των εργαζομένων Παλαιστινίων ε, στην Κοιλάδα του Ιορδάνη κλπ. είναι κάτι το θεμελιώδες και δεν μπορούμε να το αγνοούμε και να συνεχίσουμε στην Ευρώπη να καταναλώνουμε προϊόντα που ξεκινούν από τις επικισμένες περιοχές. Είναι προϊόντα που ξεκινούν από την, τον μη σεβασμό των δικαιωμάτων δικαιωμάτων των εργαζομένων. Θα ήθελα λοιπόν να επανέλθουμε και να επανεξετάσουμε το θέμα αυτό. Μετά τι διακοπέ σίγουρα θα το επανεξετάσουμε. Πρέπει κάτι να κάνει η Ευρώπη για αυτό το θέμα τη εισαγωγή γεωργικών, μεταξύ άλλων γεωργικών προϊόντων από τι επικισμένε περιοχέ. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμεί, θα το κάνουν οι πολίτε και θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπω αυτά που είδαμε με τον στολίσκο έξω από τη Γάζα. Οι πολίτε κάνουν τη δουλειά που δεν κάνουμε εμεί οι πολιτικοί και για το θέμα των ε, ε, επικισμένων περιοχών περιοχών ακριβώς το ίδιο ισχύει. Ε, ακριβώς για το θέμα της αξιοπρέπειας και της ε, ε, εισάξιας αξιοπρέπειας Ισραηλινών και Παλαιστινίων θέλω να πω ότι ζητούμε την απελευθέρωση του Γκλάτ Σαλίντ άμεσα, αλλά ζητούμε παράλληλα και την απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων εχμαλώτων που βρίσκονται στη φυλακή πριν από τις συμφωνίες του Όσλο υπάρχουν νέοι ανήλικοι που βρίσκονται στο Ισραήλ στη φυλακή και αυτό είναι απαράδεκτο. Επίσης, η ίση μεταχείριση θα πρέπει να ισχύει μεταξύ ενός ε, ευρώ Ευρωπαίου Ισραηλινού όπως ο Σιλάτ Γκαλίτ και ο Σιλάτ Αμουλιά που είναι Ευρωπαίος Παλαιστίνιος ε, εδώ και χρόνια στη φυλακή και αυτό είναι επίσης απαράδεκτο. Θέλουμε ο Σελά Αμουλή να απελευθερωθεί. Τέλος. Ανέφεραν οι συνάδελφοι τι συνέπειε του αποκλεισμού, αλλά θα ήθελα να πω ότι ο αποκλεισμό ευνοεί τη Χαμά και ε, ο αποκλεισμό είναι κάτι που είναι κατά των παιδιών, κατά των γυναικών, γιατί η βία κατά των γυναικών μέσα σε αυτή την κατάσταση καταπίεση, μέσα σε την κατάσταση του αποκλεισμού, κάνει τις γυναίκες θύμα του, του αποκλεισμού. Οι καλλιτέχνες, οι διανοούμενοι είναι θύμα του αποκλεισμού. Συναντήσαμε κάποιον καλλιτέχνη και οι καλλιτέχνες πραγματικά είναι ιδιαίτερα καταπιεσμένοι στη Γάζα. Ο αποκλεισμός είναι κάτι που είναι ενάντια σε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να λάβει μέτρα η Ευρώπη το συντομότερο δυνατόν για να σταματήσει αυτός ο αποκλεισμό και τέλος θα ήθελα να πω την κρίμα που λείπει ο Πρόεδρος, διότι αν υπάρχουν κάποιες ε, διαφωνίες ε, όσον αφορά ε, τη διοργάνωση μιας προσπάθειας. Είναι κάτι το οποίο είναι λογικό μέσα σε μια δημοκρατική διαδικασία, αλλά θα, θα έπρεπε να είναι παρόν για να ε, ακούσει τα σχόλια, για να ακούσει τη συζήτηση, γιατί ακριβώς έτσι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους να καταλήξουν σε συμφωνία και ειρήνη μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Κύριος Βάγκε. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω κι εγώ ε, την, τις ευχαριστίες μου προς τον ε, κύριο Παντσέρη. Εκτιμώ ιδιαίτερα την ε, παρουσίαση που μας έκανε για την επίσκεψή μας. Έχουμε συζητήσει τις τελευταίες εβδομάδες τα θέματα αυτά και τα συμπεράσματα στα οποία μπορούμε να καταλήξουμε μετά την επίσκεψή μας και δεν χρειάζεται να επαναλάβω και εγώ αυτά που είπαν άλλοι συνάδελφοι. Η επίσκεψη έγινε την κατάλληλη στιγμή. Δείχνει την, ε, το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου και το πώς ε, θέλουμε ε, να συμμετέχουμε στις προσπάθειες αυτές υποστήριξης των πολιτών και των φορέων, γιατί είναι ένα από τα καυτά θέματα της διεθνούς πολιτικής. Και εγώ θεωρώ ότι είναι κρίμα που ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, ΑΦΕΤ ε, δεν ε, έχει το ηθικό ανάστημα να συμμετάσχει σε αυτές τις συζητήσεις. Είναι κάτι στο οποίο αναφέρθηκαν και οι Ισραηλινές εφημερίδες, ότι η αντιπροσωπεία έκανε ε, προπαγάνδα κατά του Ισραήλ. Και πιστεύω ότι θα έπρεπε ε, να φροντίσουμε να αποσυρθούν αυτά τα οποία ε, δηλώνονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Και τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε ακούσει τα σχόλια που έχουν γίνει και τις παρατηρήσεις του Πρωθυπουργού κυρίου Φαγιάτ και της ΟΝΡΑ. έχω την εντύπωση ότι η λύση των δύο κρατών που ανέφερε ο κύριος Πέτερινγκ ως σημαντικό στόχο τον οποίο υποστηρίζουμε, είναι μια λύση που φαίνεται σχεδόν ε, μη πιστευτή με βάση αυτά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στη Δυτική Όχθη. Όσον αφορά την υποδομή, όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού, σαφώς βλέπουμε ότι δεν παρέχονται ίσα δικαιώματα στους Παλαιστινίους. Οι Ισραηλινοί ετοιμάζουν ε, τρία νομοσχέδια που αφορούν στην οργάνωση της ε, κοινωνίας των πολιτών και αυτό θα, αυτά θα δυσκολέψουν ιδιαίτερα την ε, οργάνωση των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νέιτς, ευχαριστώ συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που μας ανέφεραν ε, τα συμπεράσματα της επίσκεψης της αποστολής αυτής. Δυστυχώς δεν μπόρεσα για οικογενειακούς λόγους να συμμετάσω εγώ, αλλά ε, προηγήθηκαν τα επεισόδια που γνωρίζουμε και τα οποία συζητήσαμε επί μακρόν σε έκτακτη σύνοδο του διευρυμένου Προεδρείου της ε, Επιτροπής μας, την οποία είχα συγκαλέσει εγώ ε, με υποστήριξη όλων των υπολείπων πολιτικών ομάδων στο Στρασβούργο πριν από δύο συνόδους. Θα ήθελα να θυμίσω στους συναδέλφους μια δήλωση που είχε γίνει ενώπιον της Επιτροπής μας από το μόνιμο αντιπρόσωπο του Ισραήλ ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν συζητήσαμε ε, την επίθεση στην Ιωπομπή που κατευθυνόταν προς τη Γάζα ε, και είχε στόχο να προσπαθήσει να σπάσει τον αποκλεισμό. Είπε λοιπόν ο μόνιμος εκπρόσωπος του Ισραήλ ότι όντως το Ισραήλ αντιτίθεται σε επισκέψεις βουλευτών και άλλων ε, προσωπικότητων στη Γάζα, διότι, και νομίζω το παραθέτω από μνήμης, αλλά νομίζω ότι ε, σωστά το λέω, ότι τέτοιου είδους επισκέψεις, λέει, νομιμοποιούν την κατάσταση στη Γάζα. Το καθεστώς. Δηλαδή, και ε, μόνο πηγαίνοντας εκεί εμείς, στα μάτια της Ισραηλινής κυβέρνησης, την οποία υποθέτω εδώ προσωπεί ο μόνιμος αντιπρόσωπος, ή αν μη τι άλλο τη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι αυτή. Το είπε εδώ στην Επιτροπή μας, ενώπιόν μας. Ότι τέτοιου είδους επισκέψεις θεωρούνται όχι απλώς άστοχες, αλλά και τελείως ανεπιθύμητες και θα πρέπει όσο γίνεται περισσότερο να αντιταχθούμε και να τις αποτρέπουμε, διότι ε, αυτό προσδίδει νομιμότητα στη κατάσταση στη Γάζα. Ελπίζω η ελαφρά αλλαγή ε, στάσης που ανέφερε η Βερονίκη το Ισραήλ και που λίγο, τόσο λίγο ε, χαλαρώνει τον αποκλεισμό να σηματοδοτεί και άλλη αλλαγή. Αλλά νομίζω αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και να μην το ξεχνάμε. Να πιστεύουμε δηλαδή ότι μπορούμε να εξευμενήσουμε το ε, Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κάνοντας δεν ξέρω εγώ τι, είναι χήμερα και αυταπάτη. Δεν ήταν όλοι παρόντες, γι' αυτό τα ξαναλέω όταν είχε έρθει ο πρόσωπος στην Επιτροπή. Είναι βαρισίμαντη αυτή η δήλωση. Πολύ. Και δυστυχώς πολύ κακός ιονός για το μέλλον. Ε, ο κύριος Μαύρο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τους συναδέλφους που μας ενημέρωσαν για τα της στη Γάζα, νομίζω ότι σωστά παρουσίασαν τα πράγματα, πονώντα όχι μόνο ποιο είναι το δράμα που ζουν οι άνθρωποι εκεί, αλλά όπως έκανε ο κ. Πέτερινγκ, υπογραμμίζοντας τον τελικό σκοπό της επισκέψής μας, που είναι να καταλήξουμε στη λύση δύο λαοί, δύο κράτη. Αλλά για λόγους ρεαλισμού, διερωτώ με, όσοι είναι υπέρ αυτή τη λύση. Δύο, λέει, δύο κράτη έχουν αυξηθεί ή έχουν μειωθεί. Και συγκεκριμένα έχουν αυξηθεί ή μειωθεί τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Παλαιστίνη. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι και στι δύο περιπτώσει έχουν μειωθεί οι υπέρμαχοι αυτή τη λύση. Και στο εσωτερικό τη Ισραηλινής κυβέρνηση και δεδομένων των δηλώσεων των επικεφαλής της Χαμάς. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ποια είναι η δική μας ευθύνη. Επίσης, ο πρόεδρος Πέτερινγκ μίλησε για την στήριξη που θέλουμε να προσδώσουμε στον Αμερικανό πρόεδρο ώστε να φέρει στο σωστό δρόμο την διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Αλλά και εδώ θα ήθελα για λόγους ρεαλισμού να κάνω μια παρατήρηση. Όλοι όσοι έκαναν δηλώσεις και πιο συγκεκριμένα το τάγμα στρατιωτών από την Ιταλία στα νότια του Λιβάνου και οι δηλώσεις λοιπόν σχετικά μας δίνει την εντύπωση ότι άλλα λένε βρίσκονται επί τόπου και η Αμερικανική κυβέρνηση ασχέτως από τις προθέσεις του Πρόεδρου Ομπάμα δεν σημαίνει ότι πράττει τα ίδια μέσω του προσώπου της ε, Υπουργού Κλίντον. Έτσι λοιπόν, η επιρροή που ασκείται από συγκεκριμένε κατευθύνσεις προς την Αμερικανική κυβέρνηση είναι ισχυρή. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και νομίζω, και εδώ θα καταλήξω, και θα συμφωνήσω με το σημείο που τόνισε και ο συνάδελφο Παντέρη. Νομίζω λοιπόν ότι οφείλουμε, έχουμε το καθήκον μέσω των μέσων που έχουμε προβλέψει, να δώσουμε έμφαση στην ομάδα εργασία για τη Μέση Ανατολή, όπου προεδρεύει ο κ. Πέτερη, και εκεί να φροντίσουμε να σκεφτούμε τα πράγματα με γνώμονα τον, την πραγματικότητα, την αλήθεια. Δηλαδή, τον πραγματικό μας σκοπό, δύο, λέει, δύο κράτη χθες, ο ε, πρέσβη του Ιράκ μα είπε με τρόπο πολύ ειλικρινή και συνεπή ότι οι υποθέσει τη χώρα του και τα προβλήματα τη χώρα του σχετίζονται με το γεγονό ότι άλλοι παράγοντε του Ιρακού κόλπου, η Σαουδική Αραβία και το Ιράν, παρεμβαίνουν για δικού του σκοπού εξουσία. Αυτό λοιπόν δεν είναι δυνατόν να, μην, να ισχύει για το Ιράκ και να μην ισχύει για το Ισραήλ ή για την Παλαιστίνη. Θα πρέπει να τα έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μα ότι όλοι οι παράγοντε δρούν ταυτόχρονα σε αυτή την περιοχή. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου σημαίνει αυτό για τι συνέπειε που προκαλούνται. Γιατί η δική μα η συνεισφορά θα πρέπει να είναι μια συνεισφορά στην κατεύθυνση τη αλήθεια, τη πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να κάνουμε και όχι να χάνουμε χρόνο με εσωτερικέ διακλονικίε. Ο κύριο Αγκουράκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη, νομίζω ότι πρέπει ακόμα περισσότερο να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό δεν είναι θέμα ίσων αποστάσεων. Ο Παλαιστινιακός λαός είναι εκείνος που υποφέρει, εκείνος είναι που δεν έχει κράτος. Εάν θέλουμε να υλοποιηθεί αυτό που λέμε δύο κράτη, δύο λαοί, πρέπει να ενισχύσουμε αυτό που είναι πιο αδύνατος και επίσης να θυμίσω ότι ο Παλαιστινιακός λαός υποφέρει γιατί ε, βρίσκεται υποκατοχή. Άρα δεν μπορεί η κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ να είναι το ίδιο πράγμα με την αντίδραση ενός λαού που βρίσκεται υποκατοχή. Το δεύτερο που ήθελα να σημειώσω είναι το εξή παρά την απαράδεκτη επίθεση την οποία όλοι την καταδικάσαμε του Ισραήλ ενάντια στην, ε, ε, στον στολίσκο που ήθελε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας είδαμε όλοι ότι δεν ενθουσιάστηκε ή μάλλον είδαμε όλοι ότι δεν εντυπωσιάστηκε και πάρα πολύ η Ισραηλινή κυβέρνηση. Είδα τον Πρωθυπουργό της χώρας να έχει το θράσος, να λέει ότι η χώρα του έχει ανταποκριθεί στο διεθνές αίτημα υπάρχει Διεθνή Επιτροπή λέει, που εξετάζει το συμβάν. Και πρέπει να σα πω κύριε Πρόεδρε ότι νομίζω ότι στη στάση αυτή τη κυβέρνηση του Ισραήλ έχει συμβάλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των επίσημων τοποθετήσεων και τη κυρίας Άστον και του ε, Συμβουλίου αμέσως μετά τα γεγονότα που περιορίστηκε σε μια πολύ χλιαρή τοποθέτηση και δεν πήρε κανένα αντίμετρο στις σχέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ισραήλ. Παραδείγματος χάρη θα μπορούσε να είχε ε, απαγορευτεί, να, να είχε παγώσει η στρατιωτική συνεργασία με το κράτος αυτό το επιθετικό. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι εμεί έχουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική τη απέναντι στο Ισραήλ, ε, αν θέλουμε να συμβάλλουμε ακόμα πιο πολύ ε, στην επίλυση του ζητήματο. Και ένα τελευταίο ζήτημα. Νομίζω ότι πρέπει ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απευθυνθεί και να στηρίξει ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω σε τι βαθμό το κάνει, δεν άκουσα τίποτα, αλλά πρέπει να στηρίξουμε και εκείνε τι δυνάμει στο εσωτερικό του Ισραήλ, όπω είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπω είναι η Χαντά, όπω είναι το αντιπολεμικό κίνημα το οποίο αγωνίζεται για μια επίλυση του προβλήματος για δύο ανεξάρτητα κράτη, για την ειρήνη και οι οποίοι άνθρωποι και δυνάμεις υποφέρουν πάρα πολύ από, το καταπιεστικό, ε, από τα καταπιεστικά μέτρα της κυβέρνησης του Ισραήλ που στοχεύουν ακόμα και μέλη της Κνεσέτα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you, Mr. Weber, please. Weber. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας Ντεκάιζερ, αν τα 20 εκατομμύρια που προβλέπονται, εφόσον το Κοινοβούλιο δώσει την έγκρισή του και επιτρέψει να μεταφερθούν 40 εκατομμύρια, η πρόταση που έχει υποβληθεί νομίζω το πρωί μόλι του συναδέλφου τη Επιτροπή Προπολογισμών, το ίμιση των 20 εκατομμυρίων στόχο έχει να ε, ενισχύσει τον προπολογισμό που προβλέπουμε. Τώρα, αν είναι επαρκή αυτά τα κονδύλια. Κοιτάξτε, το έλλειμμα της Ούρα για το 2010 και εφόσον ο προσωρινός προπολογισμό της κατά 100 εκατομμύρια δολάρια μειώθηκε ήδη, φτάνει τα 75 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την αφαίρεση των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Για να αντιμετωπίσει τις δαπάνες της, 85% των οποίων καλύπτουν τους μισθούς των εργαζομένων της ΟΥΡΑ. Αυτά τα έξοδα δεν μπορούν να μειωθούν, εκτός αν απολυθούν άνθρωποι. Αυτά τα 20 εκατομμύρια προφανώς θα επιτρέψουν απλώς να καλυφθεί λίγο το έλλειμμα των 75 ε, εκατομμυρίων κατά το 1 τρίτο, κάτι λιγότερο. Έτσι λοιπόν θα απομένουν κάποια εκατομμύρια ευρώ στην Ούνρα για να καλύψει κάποια από αυτό που έχει αναλάβει με ένα προπολογισμό ήδη περιορισμένο. Κατά 100 εκατομμύρια δολάρια μειωμένο όπω υπάρχει Δεν είναι αρκετά βεβαίω. Αλλά τουλάχιστον θα καλυφθούν κάποιε άμεσε ανάγκε τη ΟΥΡΑ και όπω τι εξέφρασε στην επιστολή που απίθυνε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπω γνωρίζετε με το αντίγραφο που λάβατε. Και εκεί ζητήθηκαν και τα 20 εκατομμύρια. Έτσι Νομίζω ότι η Επιτροπή θα επανέλθει στο Κοινοβούλιο ενώπιον τη αρχή προπολογισμού τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο για να επαληθεύσουμε κατά πόσον οι ανάγκε τη ΟΥΝΡΑ είναι πολύ σοβαρέ ακόμη και αν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τι καλύψουμε εν μέρη από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση και αν οι ανάγκε που εντόπισε ο Πρωθυπουργό Φαγιάντ και που μίλησε σε εσά και του συναδέλφου σα χθε μπορούν να καλυφθούν από τα 40 εκατομμύρια που θα διαθέσουμε εφόσον και εσείς δώσετε τη δική σας έγκριση. Τώρα, η κατάσταση στην ε, Γάζα. Δεν φαντάζομαι να χρειάζεται να κάνω κι εγώ καταληκτικά σχόλια, το είπατε όλοι. Είναι πολύ θλιβερή. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπων που βρίσκονται σε μια μεγάλη φυλακή, δεν μπορούν να βγουν. Ούτε τη ε, αεροπορική ούτε από τη θάλασσα, ούτε από την ξηρά. Αυτό θα μπορούσε να κρατήσει Ήδη έχει κρατήσει πολύ. Υπερβολικά πολύ ο αποκλεισμό. Τώρα, αν είναι προφανώ δημοκρατικό, εγώ δεν έχω άποψη. Εσεί θα το κρίνετε. Σω είναι μια δημοκρατία ρωμαϊκού τύπου. Οι πολίτε ε, έχουν κάποια δικαιώματα και σκλάβει κανένα. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη, ίσω. Αυτό που θεωρώ πάντω σίγουρο είναι ότι είναι απαράδεκτο να έχουμε παιδιά που δεν μπορούν να έχουν καν παιχνίδια. Γιατί απαγορεύονται και εισαγωγέ παιχνιδιών. Είναι απαράδεκτο ένα μέρο του πληθυσμού να μην μπορεί να συντηρηθεί. Ούτε να κατασκευάσει τα σπίτια που καταστράφηκαν με τα άναδομη. Και να μην πάει σχολείο. Γιατί έχουν τρία. Τρεις βάρδιες την ημέρα για να μπορέσουν να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Είναι δυστυχώς μια κατάσταση απαράδεκτη σε απόσταση 4 ώρες πτήσης από την Ευρώπη. και για ανθρώπους που μπορούσαν να πηγαίνουν στα καλύτερα πανεπιστήμια. Και πιστεύω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Η κυρία Άστον με τόλμη είπε ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη, το είπε και σε εσά και στο Συμβούλιο. Και κάτι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσει ο αποκλεισμό τη Γάζα. Γι' αυτό χρειάζονται χρήματα βέβαια. Ο Πρωθυπουργό Φαγιάντ πραγματικά βελτίωσε την κατάσταση στην Δυτική Όχθη σε οικονομικό επίπεδο και τα προγράμματα που εκτελέστηκαν με την δική μας τη στήριξη και με τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας επέτρεψαν ένα καλύτερο επίπεδο ανάπτυξη. Άρχισαν να γίνονται λοιπόν αυτά που είχε υποσχεθεί αρχικά ο κύριο Φαγιάν. Δηλαδή, μείωσε το έλλειμμα τη Παλαιστινική Αρχή, ε, μπόρεσε να αντιμετωπίσει τι οικονομικέ δυσκολίε τη δυτική όχθη εν μέρη. Από την άλλη άνοιξε η ψαλίδα. Δηλαδή η Γάζα πάει όλο και χειρότερα. Και εδώ έχουμε 1,5 εκατομμύριο Παλαιστινίου σε σχέση με τα 2,5 τη Δυτική Όχθη, που ζουν σε συνθήκε ακραία φτώχεια. Πρόεδρε, δυστυχώ, ίσω να χρειαστεί να έρθουμε και πάλι σε εσά και να ζητήσουμε συμπληρωματικά κονδύλια. Με όλα αυτά τα δεδομένα. Ο ο οποίο έχει δικαίωμα ομιλία γιατί ήταν πολύ σύντομο χθε. Ε, πάντοτε είμαι σύντομο, πρόεδρε. Δύο σύντομα ερωτήματα. Εάν οι Ισραηλοί συνεχίζουν να κατασκευάζουν, ε, να επικίζουν την δυτική όχθη και να εμποδίζουν ε, του Παλαιστινίου να μένουν στην παλιά πόλη τη Ιερουσαλήμ, δεν ε, πάβει έτσι η προοπτική τη λύση των δύο κρατών. Και αν ισχύει αυτό, εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνουμε. Thank you. Mr. Ευχαριστούμε, κύριο Παντζέρη, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Δεν θέλω να δώσω κανένα συμπέρασμα εγώ. Απλώς μια παρατήρηση και μια υπόθεση εργασίας, εάν μπορεί να γίνει. Απευθύνεται και στην Προεδρία και στην Γραμματεία. Αν θέλετε να συζητήσετε εσείς με την Προεδρία του Κοινοβουλίου, ώστε να προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα καλύτερο θεσμικό, μια καλύτερη θεσμική προβολή στην ομάδα εργασία για την Μέση Ανατολή. Διότι την ισορροπία αυτή μπορούμε να την εξεύρουμε. Και στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου θα μπορούσε να διοργανωθεί μια σημαντική διπλωματική δραστηριότητα εδώ για το όφελο τη Μέση Ανατολή. Αν μπορείτε να το σκεφτείτε. Πρόεδρος, το σημειώνουμε. Θα ξέρετε ότι στην Επιτροπή μας συμφωνούμε να χρησιμοποιηθεί το κατεπήγον ε, απόθεμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που ε, ε, με την επιστολή που έστειλε ο κ. και τον κ. Μπούζεκ. Συμφωνούμε ως προς αυτή την ανάγκη. Εγκρίνουμε λοιπόν την πρόταση. Σας ευχαριστώ. Κλείνουμε με αυτό το σημείο της ημερής διάταξης. Και τώρα η συνεδρία του Διευρυμένου Προεδρείου.